συμβολέ σα και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ε, σφαιρική προσέγγιση της Ένωσης στην μετανάστευση. Έχει υποβληθεί από την Επιτροπή ε, Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Και δίνω το λόγο στον ε, Κλοντ Μορέ. President, colleagues, The context. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτή η προφορική ερώτηση δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον νέο επίτροπό μας, επίτροπο Αβραμόπουλο, που αυτή τη στιγμή έρχεται και για να καθίσει στη θέση του. Και τον κύριο Γκότσι στο Συμβούλιο, προεδρεύοντα από την, Ιταλική Προεδρία και το Μάρεν Νόστρουμ, που θα μετατραπεί σε πρόγραμμα τρίτρων. τρίτρων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε καλά αποτελέσματα για να μην μείνουμε μόνο στα ωραία λόγια των καλών ανθρώπων αυτών που προσπαθούν να σώσουν τους μετανάστες. 3.000 πνίγηκαν το 2014 μόνο στην Ελλάδα της Μεσογείου. Σήμερα ακούσαμε τα λόγια του Αγιοτάτου Ποντίφικα που μας είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε νεκροταφείο η Μεσόγειος. Μας είπε όμως και σε ένα πολύ όριμο ε, κομμάτι της ομιλίας του ότι πρέπει να βρεθεί μια σωστή ε, πολιτική από την ε, Ένωση για να απαντήσει το πρόβλημα της μετανάστευσης με σεβασμό της αξιοπρέπειας των μεταναστών. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα αγαπητοί συνάδελφοι με το οποίο τοποθετούμεθα και διατυπώνουμε την προφορική μας ερώτηση ενώπιον του Επιτρόπου, ενώπιον του Συμβουλίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό. Πολύ άριθμα ήταν τα προφορικά ερωτήματα που έχουμε διατυπώσει. Έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά, αγαπητοί συνάδελφοι, και πρέπει να την κάνουμε. Στην τελευταία μα παράγραφα μιλούμε για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. πόσε φορέ το έχουμε συζητήσει, πόσοι τριμερεί διάλογοι έχουν γίνει, πόσα ε, νομοθετήματα, οδηγίε κανονισμοί. Αυτό που χρειάζεται είναι αλληλεγγύη. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική δράση. Και λέμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σήμερα και ιδιαίτερα κύριε Γκότση προς το Συμβούλιο, όχι την Προεδρία, γιατί στην Προεδρία έχετε ήδη τον Μαρενόστρο με 150.000 ζωές που σώθηκαν. Αλλά το Συμβούλιο δεν υλοποιεί το κοινό σύστημα ασύλου. Και άρα απευθύνομαι πρωτίστως στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Και πρέπει να αποστείλουμε και γι' αυτό χρειάστηκε να τυπωθεί σήμερα αυτό το ισχυρό ηθικό μήνυμα. Έχω λοιπόν το πρώτο τμήμα της ερώτησης προς τους δύο σας. Από το Μάρεν Όστρομ περνάμε στο τρίτο. Είναι κατάλληλο. Δεύτερον, μιλούμε για τη διεύρυνση των δραστηριότητων της Frontex. Είναι οι αρμόζουσες. Πρέπει να διατυπώσουμε το ερώτημα. Κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη όμως, εάν δεν συνεργαστούν, εάν δεν υπάρξει επιμερισμός του βάρους, τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Και μετά, ασφάλεια και νομικέ ρίζες. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να μην χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Και σε μια διάσκεψη που παρακολούθησα στο Μιλάνο, είδα ότι δεν υπήρχε πραγματική βούληση για την επαναπροώθηση ή για τον επιμερισμό του βάρους μεταξύ των κρατών μελών. Όταν λοιπόν μιλούμε για το πλαίσιο, για τα συμφραζόμενα, όπως πολλοί πράττουν εδώ, ιδιαίτερα τα μέλη, δεν πρέπει να λησμονούμε, αγαπητοί φίλοι, ότι με όλη τη λιτότητα οι χώρες που παίρνουν τους περισσότερους μετανάστες από τη Συρία και από άλλα μέρη του κόσμου, οι δέκα πρώτες χώρες η υποδοχή ε, προσφύγων δεν είναι οι προηγμένες χώρες Ευρώπης, αλλά οι, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Ούτε μία ευρωπαϊκή χώρα δεν συγκαταλέγεται σε αυτές. Πρέπει λοιπόν εμείς να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι του βάρους. Ο πρόεδρος Ιονκέρ στην εισαγωγική του τοποθέτηση μίλησε για νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να πούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ίσως όχι σήμερα, αλλά ας ξαναθυμηθούμε τι πρέπει να σημαίνει αυτό. Αγαπητοί φίλοι, ναι, κατεπήγοντα κονδύλια, ναι, κατά του, της λαθροδιακίνησης, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κέντρα υποδοχής, δεξιότητες, όλα αυτά έχουν τοτική σημασία. Ωστόσο, κύριο και κέριο σημείο, και το επισημαίνω ιδιαίτερα στην Επιτροπή και το αλλά κύριο στο Συμβούλιο είναι να υπάρχει υλοποίηση του κοινού συστήματο ασύλου. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι το αν έχει κάνει το κοινοβούλιο τη δουλειά του. Εμεί τη δουλειά μα την έχουμε κάνει. Πρέπει να κάνουμε και άλλο όμω ακόμα. Και απευθύνομαι στου συναδέλφου από την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και σε όλου του συναδέλφου του Κοινοβουλίου. Πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο πια εφαρμόστε τα εφιστάμενα νομοθετήματα. Σταματήστε τους θανάτους στη Μεσόγειο με την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Και πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στο Συμβούλιο με τους πόρους, με τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διερεύνηση των γεγονότων και να γνωρίζει και ο πολίτη ότι εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε και ότι δεν αφήνουμε να πεθαίνουν οι άνθρωποι στη Μεσόγειο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε του θανάτου αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο, είναι άλλωστε, όπως υπόθηκε και σήμερα το πρωί, μια πηξίδα ηθική. Ευχαριστώ, το λόγο έχει τώρα το Συμβούλιο. Ο, Επίτροπος, ο Υπουργός Γκότση για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μωράης που έθισε τέτοια θέματα τα οποία είναι ουσιώδη και είναι τμήμα των μεγάλων προτεραιοτήτων του εξαμένου μας ε, στη διάρκεια της Προεδρίας. Μεγάλες προτεραιότητες και το υπογραμμίζω ω Προεδρεύων με μεγάλη ικανοποίηση και το πρόγραμμα τη επιτροπή ε, Juncker που εντόπισε την ε, μετανάστευση ω άμεση προτεραιότητα και εντέταξε στο νομοθετικό πρόγραμμα ήδη του 2015 το θέμα. Να πω ότι είναι για μα μεγάλο και σημαντικό θέμα γιατί αν είναι, υπάρχει ένα θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει την αποτελεσματικότητά της ακριβώς είναι το θέμα της μετανάστευσης, εξορισμού από τη φύση της, καθώς το, θέμα, το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι διασυνοριακό. Είναι εξορισμού διασυνοριακό ζήτημα και άρα χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη κοινή απάντηση ε, και πιο θαραλέα απάντηση από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δουλέψαμε πάρα πολύ στη διάρκεια του εξαμήνου μας για να δώσουμε συγκεκριμένο νόημα σε αυτή την αρχή αυτό το άρθρο της, ε, ε, του τη συνθήκη που μιλάει για αλληλεγγύη σε θέματα μετανάστευση. Για μένα πρόκειται για μια αρχική πολιτική, πρόκειται για μια δέσμευση νομική, αλλά και για μια δέσμευση πολιτική, για την οποία πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο σε συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, την Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, που με το αίτημά του αναφέρεται στις εργασίες της Task Force για τη Μεσόγειο. Ξέρετε, συνάδελφε Μωράες, ότι ήδη ήταν 37 οι πλήρε επιχειρησιακές παρεμβάσεις της Task Force στην ε, Μεσόγειο. Θυμίζω συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε προγράμματα περιφερειακής προστασίας ε, μαζί με την ενίσχυση της δυνατότητας να φτάσει κανείς στην Ευρώπη, ε, μάλλον καταπολέμηση της σωματεμπορίας, της εποπτείας των συνόρων για να βοηθήσουμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε τους ναυαγούς στη Μεσόγειο, μέτρα στήριξη στα κράτη-μέλη που ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Αυτά όλα τα έχει δουλέψει η Task Force, τακτικά αναφέρεται δε στο Συμβούλιο και σας επιβεβαιώνω ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε δώσει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν με τη σημερινή κατάσταση. Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι και συμμεριζόμαστε τα όσα εσείς αναφέρατε Και εμεί λέμε πω η Μεσόγειο δεν μπορεί να είναι νεκροταφείο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ε, το νεκροταφείο ε, τη ε, Ευρωπαϊκή Αδιαφορία. Γι' αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο με αλληλεγγύη για να θέσουμε γρήγορα σε εφαρμογή αυτό το συνεργατικό πρόγραμμα που τελικά κρίνθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στι 10 Οκτωβρίου. Στα πορίσματα λέει ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τι μεταναστευτικέ ροές με στρατηγικό τρόπο και για να δώσουμε συγκεκριμένε απαντήσει στη μεταναστευτική πίεση γύρω από τρει βασικού προσανατολισμού, τρει βασικού τομεί πέρα από αυτού που εμεί είχαμε εντοπίσει ω προτεραιότητα ε, στη διάρκεια του εξαμήνου. Δηλαδή ενισχυμένη διαχείριση των εξωτερικών συνέωρων που επιτέλου μετά από χρόνια δουλειά και μετά από χρόνια πολύ σοβαρών ευθυνών που έχει αναλάβει η Ευρώπη στην απόθεση αυτή τη αρχή, τελικά πέρασε η αρχή ότι τα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση δεν είναι ιταλικά ή πολωνικά ή ελληνικά ή ισπανικά σύνορα. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινά σύνορα και εφόσον πρόκειται περί κοινών σύνορων θα πρέπει να υπάρχει και κοινή προσέγγιση, κοινέ πρωτοβουλίες. Από αυτό εξάλλου απορρέει και η επιχείρηση τρίτονα που θυμήσατε. Ε, βέβαια αυτό δεν αρκεί, θα πρέπει αυτό να συνοδευτεί από μια δράση πολύ πιο επιχειρησιακή και αποτελεσματική, με συνεργασία με τι τρεις χώρε, διάλογο με τι χώρε προέλευση και διέλευση των μεταναστών. Ε, με γεωγραφικό, σε γεωγραφικό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε τη Βόρεια Αφρική, αλλά οι εταιρικέ σχέσει για την κινητικότητα θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικέ, να συνδεθούν περισσότερο με την οικονομική και την εμπορική συνεργασία. Θα πρέπει να επεκταθεί και στην Αφρική κάτω από την ε, νοτίω της ε, Σαχάρα, αλλά και με τι χώρε όπου έχουμε αναλάβει δέσμευση και να επεκταθεί και στο κέρα τη Αφρική. Αυτέ είναι οι περιοχέ γύρω από τι οποίε θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η προσέγγιση. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει αυτό, να, κάνει, να σημάνει τη διαφορά. Υπάρχουν πολλά να γίνουν, γιατί μάλιστα οι ε, πρώτε εμπειρίε από την εταιρική σχέση για την κινητικότητα δεν είναι ικανοποιητικέ. Το πρέπει να το πούμε στην εδώ, να κάνουμε περισσότερα ώστε να πείσουμε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης να δεσμευτούν, να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τρόπο απτό, να συνεργαστούν μαζί μας στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και έπειτα υπάρχει ο τρίτος τομέας που πρέπει να θυμίσουμε, να, στη, να στηρίξουμε πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, κοινό σύστημα ασύλου στην πράξη, η Προεδρία ε, δεν μπορεί και ούτε μπορεί να μπει στις, στις ε, παρατηρήσεις που κάνατε εσείς γιατί αφορούν διάφορες ε, διαδικασίες κατά παράβαση. Μπορεί να υπάρχουν όντως απέναντι στα κράτη-μέλη, έναντι μάλλον των κρατών μελών, αλλά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Να σας πω μόνο το εξής. Βήματα μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στη διάρκεια του εξαμήνου μας. Υπάρχουν διάφορα ε, υπάρχουν πολλές κοινέ ρυθμίσεις, υπάρχει μια περιορισμένη δυνατότητα εξαιρέσεων, υπάρχουν βήματα μπροστά που έγιναν, αν σκεφτεί κανείς και το νέο κανονισμό στο εσωτερικό του συστήματος του Δουβλίνου, που ως Προεδρία θεωρούμε πως εν μέρη είναι ακατάλληλο. Δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, αλλά εμείς θεωρούμε πως είναι εν μέρει ανεπαρκές για να απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις, αλλά υπάρχει κάποιο περιθώριο ευελιξίας ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό μέσα στο σοβαρό θέμα της μετανάστευσης, που είναι το θέμα των μη συνοδευόμενων ανηλίκων όπου οι κανόνες μας επιτρέπουν να κάνουμε πολλά περισσότερα, όπως έχουμε και το νέο μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Σαφώς ε, στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ε, ε, παγιοποίηση και στην εδραίωση αυτού του συστήματος που υπάρχει καθώς και στη ρύθμιση τη διοικητική ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα κοινό για το άσυλο και έπειτα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια μηδέα εμπιστοσύνη γιατί τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αφήσαν Αφέθηκαν κάποια κράτη να αντιμετωπίσουν στην ουσία μόνα τους ένα μαζικό φαινόμενο που μας αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Υπήρξε λοιπόν απουσία αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κρατημέλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε για το θέμα των συνόρων, για το θέμα των τριτοχωρών, αλλά και για το θέμα καλύτερη διαχείριση Ενό ε, καλύτερου συστήματο ασύλου. Τα κρατημέλη πρέπει να βελτιώσουν τα εθνικά του συστήματα για το άσυλο, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη προπόθεση ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια πραγματική νέα πολιτική μετανάστευση. Α το σκεφτούμε αυτό, ότι ω Προεδρία στη διάρκεια του εξαμήνου μα, εμεί προτείναμε την αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση, επί το οποίο δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, αλλά που είναι σίγουρα μια από τι απαντήσει για να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα στο οποίο αναφερόμουν, που χρειάζεται όμω το συγκεκριμένη προπόθεση να ισχύσει, να επαστρέψουμε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εφόσον δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να ασκηθεί αυτή η πολιτική μετα... κοινή πολιτική μετανάστευση που μπορεί και πρέπει να αναπτύξει οπωσδήποτε η Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Δίνω τώρα το λόγο στον Επίτροπο, κύριο Αβραμόπουλο. Παρακαλώ, μέρος Επιτροπής. Uh, thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μετανάστευση ήταν πάντα στο χαρτοφυλάκιο των εσωτερικών υποθέσεων. Αλλά ποτέ δεν συμπεριλαμβανόταν στον τίτλο, στην ονομασία. Τώρα όμως ναι, περιλαμβάνεται και για συμβολικούς λόγους αλλά και για ε, ρεαλιστικούς λόγους. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στον Πρόεδρό της, τον κύριο Μωράης, διότι μου έδωσαν τη δυνατότητα σήμερα να είμαι εδώ σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω αυτά τα οποία είπε το πρωί ο Πάπας Φραγκίσκος, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. και νομίζω ότι διερμηνεύω όλων ε, την άποψη από ότι το ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψε το λάβαμε και με πλήρη σεβασμό στις παρατηρήσεις του. Πραγματικά με τιμά που έχω αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν το κρύβω. Ταυτόχρονα βέβαια γνωρίζω ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση για την ε, αντιμετώπιση του πολύ σημαντικού αυτού καθήκοντος που έχουμε ενώπιόν μας. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει έντονη, ισχυρότατη πολιτική βούληση από πλευράς μας. Τα διεξοδικά σας ερωτήματα δείχνουν πόσο πολύπλοκες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλότερες μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά μας σύνορα μετά την κρίση στα Βαλκάνια. Απαιτείται γι' αυτό μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς και την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας μεταξύ αυτών. Πρέπει να αποκαταστήσουμε, να οικοδομήσουμε μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτούς, αυτές τις προκλήσεις με επιτυχία. Εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών αλλά και των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Και σίγουρα πρέπει να υπάρξει και ένας επιμερασμό ε, των ευθυνών, διότι αυτό είναι ακρογωνιό λήθος, αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό σύστημα μετανάστευση και ασύλου με κοινά πρότυπα, κανόνες ε, και δικαιώματα όμως για τους μετανάστες. Ε, πολλά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για την αλληλεγγύη, για το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη αυτά. Έχουμε την οικονομική αλληλεγγύη, υποστηρικτικά μέτρα και την υποστήριξη παρέχει ε, και το Frontex και ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Υποστήριξη του Ασύλου και η σχετική εθνική φορήση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει το λιθαράκι της και σίγουρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έχουμε τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, έχουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει και το άρθρο 33 του κανονισμού Δουβλίνο 3. Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους. Πρέπει όμως και να τα αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αλληλεγγύη συμβαδίζει με την ευθύνη, την υπευθυνότητα. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να οικειοποιηθούν πλήρως αυτή τη διαδικασία για να λειτουργήσει όσο πιο καλά μπορεί αυτό το σύστημα. Η πλήρης αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ την υλοποίηση από τα κράτη-μέλη και θα στηρίζει και τις προσπάθειές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και στην πρακτική συνεργασία, μέσω του ΕΑΖΟ κυρίως. Βέβαια, βασιζόμαστε και στην ε, συνεχή υποστήριξη που μας παρέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή διεθνείς εταίροι όπως ε, είναι η πατιαρμοστία του για τους πρόσφυγες. Έχουμε κανόνες που ισχύουν, όπως το Δουβλίνο 3. Αλλά από τον Ιούλιο θα ε, ισχύσει νέες ρυθμίσεις. Δεν ε, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα ασύλου, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι επίγον αυτό. Όμως, μεσοπρόθεσμα, ε, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μπορεί να γίνει, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Η διακίνηση, το λαθρεμπόριο έχουν και ένα στοιχεία μεταξύ τους, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά ε, ποινικά δικήματα. Και γι' αυτό πρέπει οι απαντήσεις μας να είναι προσαρμοσμένες στο καθένα ξεχωριστά για την ε, πορεία ανθρώπινων ε, όντων, ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι στο επίκεντρο της δράσης μας και εντάσσεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να προστατεύσουμε όλα τα θύματα και θα πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση ε, για τους ε, διακινητές, ε, ποινική απάντηση. Θα προτείνουμε λοιπόν δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της διακίνησης. Η πρόληψη είναι επίσης κλειδί. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να αναλάβουν δομική δράση για να μειώσουν ε, όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για την ε, ποινικοποίηση των ε, εργαζομένων, είτε για την τιμωρία αυτών που χρησιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες γνώση τους. Θα πρέπει να είμαστε πιο επιτυχείς στην ανταπόκρισή μας σε αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει να πάψουν αυτές οι εγκληματικές ενέργειες. Θα πρέπει να διωχθούν και να τιμωρηθούν πιο αυστηρά οι δράστες. Έχουμε ένα σχέδιο ε, στο μυαλό μας ε, για την καταπολέμηση ε, της διακίνησης και αυτό θα εστιάζεται και στην ε, εξάρθρωση αυτών των δικτύων και στην ενίσχυση της διάδοσης ε, και ανταλής πληροφοριών και στην αύξηση των δυνατοτήτων μας ε, στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της δίωξης. Θέλουμε ενημερωτικές εκστρατείε για τους κινδύνους που ενέχει η διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε βελτιωμένη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Η απάντηση στις μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορα και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου για της διακίνησης συνεπάγονται και έναν πιο ισχυρό ρόλο για την Frontex. Θα πρέπει να διευρύνουν ε, τα κράτη-μέλη της της Frontex, θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά με την υπηρεσία αυτή. Μόνο τα κράτη-μέλη έχουν ε, το και στη διάθεσή τους και τα άλλα απαραίτητα μέσα. Σε ό,τι αφορά το τρίτον, την κοινή αυτή επιχείρηση, ξέρετε ότι Ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος η επιχείρηση τρίτων και θα, εξελιχθεί, θα εξαρτηθεί το μέλλον της από το πώς θα λειτουργήσει και τι αποτελέσματα θα έχει. Θα παρακολουθούμε ε, βέβαια, αλλά η υπηρεσία και τα κράτη-μέλη θα έχουν την ε, τελική ευθύνη. Το κόστος υπολογίζεται σε 2,9 εκατομμύρια το μήνα. Για τη δρομολόγηση και χρηματοδότησή του βράχει πρόθεσμα έγινε μια αναδιανομή πόρων από την υπηρεσία και παρήχαμε και εμείς με άμεση μεταφορά πίστοσης 3,9 εκατομμύρια από το Ταμείο Στερικής Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει τροπολογία, να έχουμε δηλαδή ένα αποθεματικό 20 εκατομμυρίων που θα προσθεθεί στο προπολογισμό της Frontex το 2015. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση και θα δούμε τι θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο και τι θα αποφασίσει και το Συμβούλιο. Με το άσυλο δείχνουμε ε, αλληλεγγύη ε, και προσωπικός τρίτων χωρών. Ελαφρύνουμε κάπως το βάρος ε, ε, των χωρών υποδοχής. Τώρα, τι θα γίνει με τη μετεγκατάσταση και πόσα άτομα. Ε, αυτό είναι αρμοδιότητα των μελών. Εμείς θα ενθαρρύνουμε ε, την αύξηση των ποσοστώσεων. Ή τέλο πάντων όσοι δεν το κάνουν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία τη ε, μετεγκατάσταση. Εδώ όμως κάτι είναι εκτός ισορροπία. Τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν τις περισσότερες ε, αυθόρμητες αιτήσει ασύλου είναι και αυτέ που δέχονται τις περισσότερου πρόσφυγες. Και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ω Κομισιόν αυτό το ζήτημα. Χθε. οι υπηρεσίε μου είχαν ε, μια πρώτη συζήτηση διερευνητική με τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο ενός μηχανισμού κατανομής ή επιμερισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη ε, και προσιλωμένη στο να διερευνήσει και νέες επιλογές και νέες οδούς για την κοινή προσέγγιση έκδοσης ανθρωπιστικών θεωρήσεων ενδεχομένως για όσους έρχονται στην Ευρώπη και ε, ζητούν προστασία. Αυτό συζητήθηκε και στη χθεσινή συνάντηση. Αντιλαμβάνομαι ότι παραμένει άκρος λεπτό το ζήτημα αυτό σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Για προφανείς δημογραφικούς και οικονομικούς λόγους, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ε, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τη γύρανση ε, του πληθυσμού της Υπήρου μα. Συνεργαζόμαστε στενά με τους, κοινωνικού με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις. Θα δούμε τι διστάμενες πολιτικές έχουμε την μπλε κάρτα για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ελκυστική και αποτελεσματική την ισχύουσα διαδικασία και κατάσταση. Η απάντηση, κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκεται και στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Πρέπει να βελτιώσουμε τους δεσμούς μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασύνδεσή τους και να δώσουμε έμφαση στην υιοθέτηση μια μακρόπνοη πολιτική που θα αντιμετωπίζει τι βαθύτερες αιτίε ε, τη μετανάστευση. Υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο να ανταποκρινόμαστε σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη και έκτακτα περιστατικά, αλλά να έχουμε μια δομημένη προσέγγιση για μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια προσέγγιση που θα αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική σταθερότητα, την ανάπτυξη, την ασφάλεια, όλα αυτά να αντιμετωπίζονται ως ένα σύνολο. Να έχουμε τα κατάλληλα επιχειρησιακά και πολιτικά μέσα προς αυτό. Θέματα όπως η μετανάστευση, το άσυλο, διαχείριση κρίσεων, τροπιστική βοήθεια, ανάπτυξη, εμπόριο, εκδημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπίζονται συνολικά και με έναν τρόπο συνεκτικό και συνεπή και θα πρέπει η μετανάστευση να ενταχθεί ε, ως θέμα στι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανταπτυξιακή συνεργασία, στην πολιτική ασφάλεια. Κάτι άλλο το οποίο είναι αναγκαίο είναι να είμαστε υποστηρικτικοί αλλά και αξιόπιστοι. Να, στηριζώ, να υποστηρίζουμε τις ε, χώρε εταίρου για να διχειρίζονται καλύτερα τα σύνορά του. Θέλουμε επίση να βελτιώσουμε την ε, προστασία, τι δυνατότητε υποδοχή για να βοηθήσουμε τι χώρε να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις. Τερικές σχέσεις κινητικότητας ε, βοηθούν στην εμβάθυνση και στην ε, δημιουργία ε, των θετικών συνθήκων διαλόγου. Έχουμε το Μαρόκο, την Τινησία, την Ιορδανία, με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Μακροπρόθεσμα η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση στην πηγή είναι η καλύτερη επένδυση. Στόχος μου είναι να συνεργαστώ με την ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη και να συνεργαστώ και με τους συναδέλφους μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τον Αρμόδιο για την ε, Πολιτική Γειτονία, ε, τον Αρμόδιο για την Ανάπτυξη και την Ευρωπιστική Βοήθεια. Άλλωστε αυτό ορίζεται και στην εντολή που μας έδωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρχομαι τέλος στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο του μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εκπονεί πρωτοβουλίες ε, ύψος 53 εκατομμυρίων περίπου ευρώ για την μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Από αυτά τα κονδύλια, τα 14 περίπου εκατομμύρια ευρώ θα υποστηρίξουν ε, την καταπολέμηση διακίνηση λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης. 17 εκατομμύρια ευρώ απ' την άλλη θα δοθούν για δράσεις που θα αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, και το πρόγραμμα προστασίας για τους πρόσφυγες στην Μέση Ανατολή, τις Βορειοαφρικανική χώρες και το κέρα της Αφρικής. Το, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας έχει ένα προπολογισμό 60 δις για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και τις ε, συναφείς παρεμβάσεις στις χώρες της Μεσογείου. Επίσης, έχουμε και 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διατέθηκαν επιπλέον το 2014 για να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα, στην κρίση θα τη χαρακτηρίσω με τους Σύρους πρόσφυγες. Έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτού, οι χώρες της Ένωσης και Σέγγεν θα λάβουν πάνω από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στο πλαίσιο των δύο ταμείων ασύλου μετανάστευσης αφενός και εσωτερικής ασφάλειας συνόρων θεωρήσεων αφετέρου. Στην πρώτη γραμμή είναι τα κράτη-μέλη της Μεσογείου, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, που θα λάβουν με ένα μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των κονδυλίων. Συνολικά από κοινού 1,4 δις ε, σε όλη αυτή την ε, εξαετία. Τώρα, για έκτακτες περιπτώσεις, για το 2014, για όλα τα κρατημέλη μαζί, έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου ε, Ασύλου Μετανάστευσης και 6,8 εκατομμύρια για το Ταμείο που αφορά την εσωτερική ασφάλεια ε, σύνορα και βίζε και βίζες θεωρήσεις. Αγαπητοί βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με χαρά περιμένω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτέ τι προκλήσει και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι στη θέση μα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Αβραμόπουλε. Και τώρα προχωρούμε στη συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ξεπεράσει κατά 12 λεπτά τουλάχιστον το πρόγραμμά μας, γι' αυτό θα σας ε, επισημάνω ότι θα είμαι πολύ αυστηρός. Και θα δεχθώ μόνο πέντε παρεμβάσει με τη διαδικασία Κατστιά. Η κυρία Χολμάιερ όμως ξεκινάει με δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω θερμά και εσάς και την Ιταλική Προεδρία εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίω. είναι τέτοιο το μέγεθος του προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να υψέλθουν σε κάθε ζήτημα. Α, γι' αυτό το λόγο και θα επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά. Διάσωση μεταναστών. Καταρχάς, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια θερμά για τα λόγια σας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το ότι είπατε πόση πολλή δουλειά έχουμε μπροστά μας και πρέπει να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Και γι' αυτό έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που σχετίζεται με τη συνεργασία στην αντιμετώπιση του εμπορίου εις βάρος ανθρώπων. 250.000 άνθρωποι πέρασαν τη Μεσόγειο. Ο αριθμός των θανάτων υπολογίζεται σε 3.000 περίπου από την υπηρεσία μετανάστευσης. Δεν είναι όμως ε, σαφές πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έπεσαν θύματα εμπορίου. Πέθαναν λόγω αυτού του εμπορίου ανθρώπων ή έγιναν, ε, βρέθηκαν σε κατάσταση δουλείας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ακόμη και θύματα του εμπορίου οργάνων. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε καν να διανοηθούμε το μέγεθος αυτού του προβλήματος αφού δεν έχουμε στοιχεία. Είναι όλο και λιγότερες οι γυναίκες που πέφτουν θύματα ίσως του εμπορίου αυτού αλλά όλο και περισσότερα τα παιδιά που πέφτουν στα νύχια αυτών των εγκληματιών. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι οι αρχές δίωξη θα πρέπει να αναπτύξουν μια συντονισμένη συνεργασία. Μια συνεργασία που θα εμπλέκει και τρίτα κράτη και που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους εμπόρους αυτούς, αυτούς ανθρώπινων ψυχών. Να τους συλλάβει, να τους αντιμετωπίσει και επίσης να ε, διερευνήσει ταυτόχρονα τα μέσα εκείνα, τα νόμιμα, μαζί με την ε, θεώρηση διαβατηρίου για λόγους ανθρωπιστικούς, που θα επιτρέπουν την νόμιμη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να αναπτυχθεί και η συνεργασία λοιπόν, αλλά και η προστασία για τα θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάιερ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Ζίπελ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Είναι αναμφίβολα πολύ σωστό το να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη ρίζα του μετανάστευση. Μακροπρόθεσμα όμω μπορεί να φέρει μόνο αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα αμέσω. Τα μεγαλύτερα, ε, τα, τις μεγαλύτερες ροές μεταναστών δεν τις υποδέχονται τα ευρωπαϊκά κράτη, είναι αλήθεια αυτό και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει να διακινδυνεύουν και του ζωή ακόμη στον δρόμο για να βρουν γη ευρωπαϊκή και χάνουν τη ζωή τους πολύ συχνά. Πρέπει να προσφέρουμε λοιπόν προστασία από τη δίωξη, ε, από, τον πόλεμο στους ανθρώπους αυτούς. Ναι, βεβαίως λοιπόν να μην έχουμε ε, τέτοιους θανάτους, βεβαίως να μην έχουμε παράνομη μετανάστευση, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε δρόμους νόμης μετανάστευσης τότε. τότε. Είναι πολύ αυτοί οι οποίοι έρχονται ως μετανάστες. Είναι πολύ λίγα όμως τα κράτη που δέχονται μια χούφτα μεταναστών νόμιμα. Πρέπει να βρούμε λύσεις λοιπόν για τους ε, πρόσφυγες που έρχονται να στήσουν προστασία στα κράτη μας. Χρειαζόμαστε ένα καλό, μια καλή κλίδα κατανομής και επιμερισμού αυτών των ε, προσφύγων και ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες, τους. Τις ευθύνες του. Η κλίδα κατανομής, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, δεν θα πρέπει να σημάνει μόνο μείωση του φόρτου για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Σημαίνει αύξηση του φόρτου για τη Σουηδία και τη Γερμανία. Θα πρέπει δηλαδή και αυτές να συμβάλλουν μέσω μιας κλίδας κατανομής και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Χρειάζεται επίσης να αναπτυχθούν νόμιμοι δρόμοι μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Ο πρόεδρος διακόπτη. Σας ευχαριστώ κυρία Ζίπλ. 1,5 λεπτό. Ο κύριος Κέρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση της μετανάστευσης ε, είναι ε, το πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσεγγίσει τη μετανάστευση με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών υποχρεώσεων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής. Πρέπει να έχουμε μια λογική και ισορροπημένη προσέγγιση. Αυξάνονται σημαντικά οι άνθρωποι που πεθαίνουν ε, ενώ προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι παράδεκτο και μη βιώσιμο. Πρέπει να είναι κάτι η Ευρώπη το οποίο μπορεί να φτάσει κανείς. Να δεν υπάρχει απλή απάντηση. Εμείς ζητήσαμε μια καθολική προσέγγιση ολοκληρωμένη που να εξετάζει όλα τα εργαλεία που έχει στη διαθεσή της η Ένωση για να απαντήσει στην κρίση. Αυτό συμπεριλαμβάνει το να δούμε τις ευθύνε του Frontex, πώς μπορούμε να σώσουμε αυτούς που είναι ευάλωτοι και, και έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης και πνίγονται στη θάλασσα. Έχουν πέσει θύματα των σωματεμπόρων που συχνά είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσουμε τις τρίτες χώρες ε, σχηρά και αποτελεσματικά. Να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε για την επανακατάσταση και την επιστροφή. Ε, να συνεργαζόμενοι μαζί τους. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και την ανάληψη ευθυνών για την άμεση διεκπαιρέωση στην πρώτη, στην πρώτη σημείο άφηξης ε, το θέμα του ασύλου, του θέματος μάλλον του ασύλου. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε ούτε διάπλατα τις πόρτες ούτε να τις κλειδαμπαρώσουμε. Ε, και αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί να παιδευόμαστε με διάφορους λαϊκισμούς, σας βρούμε έναν πραγματικά ρεαλιστικό τρόπο για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Κέρκχοπφ. Για δύο λεπτά η κυρία Βίξτροπ. Ε, ευχαριστώ. Είναι τραγική η κατάσταση. 336 λευκά φέρετρα είδαμε μετά από την καταστροφή της Λαπεντούζας πριν από δύο χρόνια. Ξεχνάμε όμως να πούμε ότι στη Λαπεντούζα αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ε, από πνιγμό στη Μεσόγειο θάλασσα ε, φέτος είχαμε πει ότι δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν αυτά τα πράγματα και είδαμε και τον Πάπα σήμερα που μας είπε πως ποτέ πια δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Θα πρέπει η Μεσόγειος να γίνει ένα, ε, ε, ε, κοντεύει η Μεσόγειος να γίνει ένα γιγάντιο νεκροταφείο. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό, να εξασφαλίσουμε ότι θα πάψει αυτή η κατάσταση. Θα σταματήσουμε τους εμπόρους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι στα χέρια, είναι έρμεα αυτών των εμπόρων. Είναι αδύνατο να έρθουν στην Ευρώπη με νόμιμο τρόπο. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο πολιτικό ε, πρόβλημα να λύσουμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπαίνουν οι καλοί και οι σίγουροι να έχουμε τον Επίτροπο που να είναι με τη δική μας πλευρά, που δεν μιλά μόνο με το μυαλό αλλά και με την καρδιά, ε, να δοθεί ελπίδα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους πολιτικούς. Πρέπει ο νέος Επίτροπος να δουλέψει με αποφασιστικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Και τώρα έχει ερώτηση η κυρία Βάιμπερκ. Δέχεστε. Κυρία Βίξτρομ, ε, δέχεστε μια ερώτηση με μπλε κάρτα από συνάδελφο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ξέρω πως έχουμε ήδη συστήματα νομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη δεχτεί πρόσφυγες. Αλλά εσύ, Σεσίλια, πιστεύεις ε, πως πρέπει το, ο νόμος να υποχρεώνει κάποια κράτη, τα κράτη-μέλη μάλλον να δέχονται ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε, ήταν ονειρεμένη η ερώτηση αυτή. 14 χώρες ε, έχουν ανοίξει τα σύνορά τους για επανεγκατάσταση και ορισμένοι δέχονται μόλις 100 ε, ανθρώπους το χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται μόνο το 7% από όλους τους πρόσφυγες που υπάρχουν. Πιστεύω πως πραγματικά η νόμιμη μετανάστευση αλλά και σημεία επαφής ε, για τους μετανάστες, ας πούμε, στις ε, πρεσβείες μας, θα ήταν κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Ευχαριστώ. Ε, κύριε λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, δεν με ικανοποίησαν, το αντίθετο μάλιστα τα όσα είπε ο κύριος Βρωμόπουλος, με θλίβουν. Ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να βαγίσει εκτρά στην πολιτική ασύλου. Πάνω από 20.000 είναι οι άνθρωποι που ε, στα εξωτερικά σύνορα έχουν χάσει τη ζωή τους, απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να έρθουν στην Ένωση. Και πολλοί αγνοούνται και πολλοί συγγενείς αγωνιούν και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί. Χρειάζονται υποστήριξη για να βρουν τους ανθρώπους τους, να πάρουν πληροφορίες για τη μοίρα τους. Ε, είναι ε, απάνθρωπο αυτό και εκτρό ως αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη δεν είναι ανθρώπινη η ε, προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει εμείς να είμαστε πρωτοπόροι σε μια ανθρώπινη ε, δεν χρειαζόμαστε ένα τρίτο, ένα μάρε νόστουμ χρειαζόμαστε για να σώζουμε ανθρώπους, ευρωπαϊκό. Τότε μόνο είναι ανθρώπινη μια πολιτική ασύλου όπου σταματάει το Δουβλίνο, αρχίζει η ανθρωπιά. Θα πρέπει να καταργηθεί το Δουβλίνο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνε δεσμευτικέ για του πρόσφυγε, να του δώσουν αξιοπρεπεί και δίκαιε προοπτικέ. Αυτό θα πρέπει να συζητάμε, όχι το Frontex. Ε, Κυρίε και κύριοι, το δίκαιο ασύλου είναι τα σημαντικότερα που έχουμε πετύχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου εκατομμύρια ανθρώπων δεν έπαιρναν άσυλο και ήταν έρμεο στα χέρια των Ναζί. Το άσυλο είναι ένα ανθρώπινο ε, δικαίωμα αναπαλωτρίωτο το και ατομικό. Ε, αυτά θέλω να ακούσω να μου πείτε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ένστ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Κέλλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να το αγνοεί ούτε εμεί ε, ότι να πνίγονται άνθρωποι στη Μεσόγειο. Αυτοί είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από πολέμου, από διώξει, από διακρίσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πάρα πολύ συχνά πέφτουν θύματα στη ε, δράση ή την αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απίστευτα επικίνδυνο το ταξίδι που ξεκινάνε. Για ποιο? για, λόγο, γιατί δεν τους αφήνουμε άλλη επιλογή, καμία. Γιατί δεν τους αφήνουμε άλλη επιλογή, παρά μόνο να πέσουν στα χέρια των διακινητών και να τους εμπιστευτούν. Εμείς είμαστε συνένοχοι των διακινητών. Εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του κόσμου και να τον εκβιάζουν. Γιατί εμείς κλείνουμε τις θύρε προς την Ευρώπη. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιταχθούμε και να σταματήσουμε τους διακινητές, θα πρέπει να βρούμε δρόμους ασφαλείς και νόμιμους και να τους ανοίξουμε προς την Ευρώπη. Το είπε ε, ο συνάδελφος προηγουμένως, τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που λείπει μόνο είναι πολιτική βούληση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Για δύο λεπτά. Αγγέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω τον λόγο εξ ονόματος της συναδέλφου Φεράρα που απουσιάζει λόγω υγείας. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα προσπαθεί να βρει μια καλή ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία πλέον δεν είναι ε, επίγουσα αλλά ρουτίνας. Μετά από την Στοκχόλμη και το ε, Δουβλίνο ε, είχαμε εκατοντάδες νεκρών εκ των οποίων 3.000 μονάχα στη Μεσόγειο φέτος αυτό το είναι το ε, σύνορο που είναι το πιο επικίνδυνο σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της μετανάστευσης. δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε, να χτίζουμε όλο και περισσότερα φρούρια και τείχη γύρω από αυτό το φρούριο της Ευρώπης. δεν είναι δυνατόν γιατί θα απομονωθούμε ακόμα περισσότερο εμείς. Είμαστε τμήμα του βόρειου κόσμου, είμαστε τμήμα του πολιτισμένου κόσμου. Ε, δεν είναι δυνατόν εμείς να δεχτούμε ε, τέτοιου είδους διαδικασίες για αυτούς που προσπαθούν να πετύχουν άσυλο, για αυτούς που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να βρουν ε, δουλειά. Θα πρέπει να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ευρώπης. Θα πρέπει να δουλέψουμε με αυτούς που δείχνουν πραγματικά ειδικό πνεύμα αλληλεγγύης και όχι με τους διακινητές, ε, όχι με αυτούς ε, που θέλουν ε, κόσμο έτσι ώστε να τον προωθούν στην επορνεία, στο εμπόριο ναρκωτικών, στα παράνομα εμπόρια και τις εγκληματικές ενέργειες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μετανάστες που είναι συχνά πάρα πολύ νέοι, είναι μορφωμένοι άνθρωποι με καλή υγεία, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτήν την κοινωνία που τους υποδέχεται θα πρέπει να δούμε με διαφορετικό μάτι τις ε, πολιτικές ε, μετανάστευσης και θα μιλάμε πλέον όχι για μετανάστες που υποδεχόμαστε αλλά για πολίτες που εντάσσονται στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Κύριε Σαλβίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ είναι ο ναός της υποκρισίας ε, και του ρατσισμού. Ε, λέτε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε όσους μετανάστες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από την ε, πείνα. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η πείνα την οποία όχι στην Αφρική αλλά στην Ευρώπη επιβάλλουν αυτοί οι οποίοι είχαν την καλή ιδέα για το ενιαίο νόμισμα και όλες αυτές τις άλλες καλές ιδέες. Και τον πόλεμο τον οποίο ζούμε κάθε μέρα ε, η Βρετανική κυβέρνηση ε, πολύ καλά είπε ότι εγώ δεν δίνω ούτε μισό, ε, μια μισή δεκάρα για αυτούς τους διακινητές. Εμείς στην ουσία βοηθάμε τους διακινητές να πλουτίσουν. 150.000 είναι οι ε, μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στις όχθες της ε, Ιταλίας. Ελάχιστοι μεταξύ αυτών είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο ε, και τελικά χιλιάδες είναι τα ευρώ τα οποία μπαίνουν στις τσέπες των επιτιδίων. Δεν είναι δυνατόν να το συνεχίσουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραία είναι να χειροκροτήσουμε τον Πάπα Φραγκίσκο όταν μας μιλάει και σηκώνεται και φεύγει αλλά από την άλλη μεριά ε, δεν τον ακούμε όταν μας ε, λέει ότι δεν πρέπει να δίνουμε χρήματα όχι για να βοηθήσουμε τους ε, πολίτες της Ευρώπης αλλά για να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ευχαριστώ. Επιτρέπετε μία ερώτηση με μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Φερά. Που είναι... Παρακαλώ, κύριος Φέρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαλβίνη, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν συντριπτική ευθύνη σε ό,τι αφορά την αποσταθεροποίηση της Συρίας και της Λιβύης. Και έχουμε πραγματικά έκρηξη της μετανάστευσης από τη Μεσόγειο. Θα πρέπει να γίνει ήπειρος μια μηχανή παραγωγής παράτυπων μεταναστών. Ο Σαλβίνη. 500 εκατομμύρια ε, ε, πολίτες της Ευρώπης ε, υποφέρουν ε, και το ξέρουμε αυτό για τα λάθη και από τα λάθη κάποιων ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις στη Συρία έγιναν λάθη, είναι γεγονός αλλά σε τούτη εδώ την αίθουσα δήθεν λόγω της Συρίας έχουν υπάρξει κυρώσεις κατά της Ρωσίας που καμία σχέση δεν έχει με όλο αυτό και που τελικά καμία βοήθεια βοήθεια δεν παρέχουν στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Σαλβίνη για μισή λεπτό κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πέρυσι, μετά την τραγωδία της Λαμπετούζα, συμφωνήσαμε για ένα ψήφισμα σχετικά με τη μετανάστευση στη Μεσόγειο. Το κείμενο αυτό υποτίθεται θα ήταν ο δικός χάρτης και θα μας επέτρεπε μια καθολική, ολιστική λέγαμε προσέγγιση για τη μετανάσταση. Και θέλαμε να μην είναι ποτέ ξανά η Μεσόγειος η θάλασσα των πνιγμένων ελπίδων. Τα είπε και ο Άγιος Πατέρας σήμερα το πρωί. Τώρα ένα χρόνο μετά είμαστε στο ίδιο σημείο. Αλλαγή, αλλαγή που να κάνει τη διαφορά. Αν δεν γίνει αυτό ε, δεν θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ζητούμε καλύτερη συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε όλα τα διαφορετικά ε, ζητήματα και τις πτυχές του προβλήματος. Μόνο έτσι θα πρέπει συνολικά σφαιρικά να λυθεί το θέμα. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε τις δράσεις με μονομένα στοιχεία σε ένα ευχολόγιο, ε, ένα checklist που θα πρέπει ένα-ένα να το διεκπαιρεώνουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Και σας ε, καλό επιγόντως κύριε Επίτροπε και τα κράτη-μέλη να αναλάβετε συγκεκριμένη δράση στο πνεύμα της αλληλεγγύης. Και βεβαίως, εάν χρειαστεί ε, να ξαναδούμε το Δουβλίνο, ας το κάνουμε. Ε, μην κλείσουμε αυτή την πόρτα, κύριε Επίτροπε. Ας μην ε, ξανάρθουμε ε, του χρόνου τέτοιο καιρό να εκφράζουμε τη λύπη μας ότι δεν έχει γίνει τίποτα και συνεχίζουν να χάνονται ζωές. Τώρα εργαζόμαστε για ένα άλλο ψήφισμα. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε και άλλες ελπίδες, φρούδες που δεν θα τηρούμε. Το Δεκέμβριο θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Μέτσο. Ενάμιση λεπτό η κυρία Κέγκε. Signor Presidente, Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλά βήματα θετικά προς το ενιαίο άσυλο, αλλά αυτά τα βήματα δεν αρκούν απέναντι σε αυτή την μεγάλη κρίση την ε, οποία, ε, η οποία βαθαίνει όλο και περισσότερο και αφορά τις ε, χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου. Η απάντηση δεν είναι η Frontex για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. 90% των Συρίων προσφύγων λαμβάνει άσυλο. Το ίδιο θα πρέπει ε, ζητάει άσυλο. Το ίδιο ε, θα πρέπει να, είναι και, να ισχύει και για τους Αφγανούς και για τους ε, υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι εύκολο για την Ευρώπη να αντιμετωπίσει θετικά αυτά τα αιτήματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ξαναδώσουμε ελπίδα σε, αυτούς, σε αυτά τα πλήθη των απελπισμένων ανθρώπων. Γιατί μαζί με τους πρόσφυγες και τις βάρκες τους βυθίζονται και οι ελπίδες μας και βυθίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι έφτασε η στιγμή ε, να επιτύχουν εναρμόνιση ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων ε, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν, η Ευρώπη να είναι πραγματικά θεματοφύλακα των συνθήκων και να μην φοβάται να δώσει κόκκινη κάρτα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων και των νόμων. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Χαλάχου. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κατά το πρώτο χτάμινο του έτους, περίπου 120.000 παράτυποι μετανάστες πέρασαν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Εξαπλάσιος αριθμός δηλαδή από ό,τι το 2013. Η επιχείρηση Mare Nostrum αύξησε τραγικά τα νούμερα αυτά, αλλά και φυσικά και τον αριθμό των τραγωδιών και των αβαγίων. Και παρά τους κινδύνους, ο θαλάσσιος δρόμος εξακολουθεί να είναι ο πιο ελκυστικός δρόμος για τους μετανάστες. Γιατί τη στιγμή που φτάσουν, που πατήσουν στην Ευρώπη, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν μια άδεια παραμονής και θα έχουν και δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση, ακόμη και αν δεν πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, να δούμε ε, ποιες, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντε ε, του κανόνε τη δευτερογενή προστασία, τη επανένωση οικογενειακή και τα κοινωνικά επιδόματα. Θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν αξίζει να διακινδυνεύει κανεί τη ζωή του και να ε, δίνει λεφτά στου διακινητέ, γιατί δεν θα επιβραβευτούν οι προσπάθειέ του. Και μάλιστα θα πρέπει να έχουμε πανευρωπαϊκέ δράσει. Πέρυσι η Σουηδία υποδέχθηκε ε, και έλαβε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων ασύλου από την Ιταλία. Πενταπλάσιο αριθμό Γερμανία. Γερμανία. Φαίνονται οι αδυναμίες ε, του μηχανισμού του Δουβλίνου και υπονομεύει μια τέτοια κατάσταση το παραδεκτό ε, και τα θετικά στοιχεία του χώρου του Σέγγεν. Θέλουμε μια νέα στρατηγική. Η διάνοιξη νέων νομικών δρόμων προς την Ευρώπη δεν είναι λύση, γιατί η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν ε, μπορεί να αντέξει τέτοιου είδους μετανάστευση, είτε είναι αυτή παράτυπη, είτε νόμιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε Χαλαάχο. Η κυρία Γκρισμπέκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Για άλλη μια φορά εδώ στο Κοινοβούλιο ε, μοιραζόμαστε τραγικές διαπιστώσεις. Μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρών Δύο φορές ακούσαμε σήμερα το πρωί από τον Πάπα που μίλησε για νεκροταφείο στη Μεσόγειο, το νεκροταφείο της αδιαφορίας όπως είπε και ο Σάνδρο Γκόζη. Αλλά απόψε ξανά μοιραζόμαστε τις ίδιες διαπιστώσεις. Η μεταναστευτική μας πολιτική δεν λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και αυτή η ολιστική στρατηγική και σφαιρική που όλοι επιθυμούμε είναι ανάγκη. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για πολιτική βούληση. Περιμένουμε από εσά ακριβώς να προκαλέσετε ε, αυτό το momentum, να αποκτήσουν αυτή την ορμή, τη φόρα τα κράτη-μέλη, να καταλάβουν ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά και να υπάρξει εκφράση ε, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του επιμερισμού, όπως είπατε και εσείς, της αλληλεγγύης. Ε, έχω λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Στην εκπόνηση αυτής της συνολικής στρατηγικής για τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα, θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους που είναι ευάλωτα όντα τα παιδιά. Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Σπινέλη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε δύο δηλώσεις. Αυτή του Ιταλού Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία έκλεισε η Μαρενόστρουμ και μετά από ένα διάστημα, ε, ε, χάρη στην Frontex, δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα σπαταληθεί πλέον ούτε ένα ευρώ για τις θαλάσσιες διασώσεις. Ο Βρετανός Υπουργός ε, λέει ότι θα πρέπει γρήγορα να σταματήσουν οι διασώσεις στη Μεσόγειο γιατί ενθαρρύνουν τους μετανάστες. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο αυτές τις δηλώσεις γιατί ε, προϋποθέτουν ή υποθάλπτουν μάλλον ένα ενδεχόμενο έγκλημα που γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε, να προκαλούμε μαζικούς πνιγμούς δεν είναι να αφήνουμε ε, εκατοντάδες ανθρώπους ε, στην Αθήνα ε, που αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πείνας. Θα πρέπει να δώσουμε τα ευρώ έτσι ώστε να σώζονται άνθρωποι. Το ακούσαμε και σήμερα το πρωί. Εάν το Κοινοβούλιο δεν αλλάξει, κόβει ο πρόεδρος στο μικρόφωνο της κυρίας Πινέλη. Για ένα λεπτό, κυρία Σεμπάγιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, η Μεσόγειος εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο πολλών επίδοξων μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει τα σύνορά της, ενώ πολλοί προσπαθούν να τα περάσουν θεωρήσαμε ότι μια ολιστική προσέγγιση ίσως αποτρέψει τους μετανάστες από το να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά πολλοί συνεχίζουν να προσπαθούν και η Frontex ήταν η απάντησή μας και στους διακινητές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νόμιμους δρόμους και νόμιμες διόδους μετανάστευσης, γιατί αυτή η είσοδος από την Κερκόπορτα είναι τρομακτική και ας μην ξεχνούμε ότι οι περισσότεροι επίδοξοι μετανάστες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την αθλειότητα στην πατρίδα τους. Θα πρέπει λοιπόν να επιληφθούμε του θέματος αυτού και να επιβάλλουμε ένα δεσμευτικό σύστημα για όλα τα κρατημέλη που θα πρέπει να αναλαμβάνουν ε, με συλλογικό τρόπο την ευθύνη τους. Ένα λεπτό, ο κύριος Μπάτεν μετά την Αραβική Άνοιξη η ανόητη ε, εξωτερική πολιτική ε, της Βρετανίας και άλλων ήταν να υποστηρίξουν τους ε, εξεγερθέντες κατά των τυράννων. Δυστυχώς οι απελευθερωτές τους ήταν οι χειρότεροι των προηγουμένων και δυστυχώς οι κάτοικοι αυτών των χωρών τώρα φεύγουν με ό,τι μέσο μπορούν κατά κύματα. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη ρίζα του κακού και η ρίζα του κακού είναι ε, μια φονταμελεστική και εξτρεμιστική ερμηνεία της Ισλαμικής ιδεολογίας ε, που βλέπουμε το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος να την εκφράζει και οι χώρες ε, που μπορούν καλύτερα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι οι πάμπλουτες Ισλαμικές χώρες ε, του πετρελαίου, Σαουδική Αραβία κτλ. Αυτές είναι οι χώρες που θα πρέπει να τους αναλάβουν γιατί έχουν και τα μέσα να τους πληρώνουν, έχουν οι ίδιες αρχές, οι ίδιες αξίες και ίδια θρησκεία τελικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάτεν. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ τώρα ο κύριος Συναδεινός. 500 άνθρωποι από τους οποίους 25 παιδιά ξεκίνησαν απεργία πείνας χθες ζητούν από το κράτο στέγη τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εργασία. προσπαθούν να μετακινηθούν σε γειτονικέ χώρε, αλλά μόλι του συλλαμβάνουν στα σύνορα του επαναπροωθούν στη χώρα προέλευση. αυτό είναι σύνηθε φαινόμενο σε χώρε όπω η συρία το ιράκ το αφγανιστάν το πακιστάν. το συγκεκριμένο γεγονό όμω συμβαίνει στη χώρα μου την ελλάδα. οι 500 αυτοί άνθρωποι κατάγονται από τη συρία. είναι ήδη συγκεντρωμένοι έξι μέρε στην πλατεία συντάγματο στην αθήνα και χθε ξεκίνησαν απεργία πείνα έτσι έχετε καταντήσει την ελλάδα όπως και άλλες χώρες στην ευρώπη του νότου όμοια με αυτές που κατηγορείτε ότι ευθύνονται για την εμφάνιση και την άνοδο του ισλαμικού κράτους και να είστε σίγουροι ότι αν συνεχίσετε την ίδια πολιτική για την παράνομη μετανάστευση η ελλάδα και, και οι άλλες χώρες του νότου δεν θα αποτελεί πλέον το μόνο πρόβλημα. έχετε αφήσει να τοποθετήσουν εκρηκτικά στις πόρτες και τα παράθυρά σας και εσείς μέσα στο σπίτι σας μαλώνετε για το πώ θα μοιράσετε το δείπνο αυτό πετύχατε με τη συνθήκη δουβλίνο 2. καταργήστε την. η ασφάλεια των συνόρων και η σταθερότητα στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή ενώσεως πρέπει να είναι το μεγαλύτερο μέλημα. η ευρωπαϊκή ένωση έχει την οικονομική δύναμη. Α τη χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει τους παράνομους μετανάστε. Α αντιμετωπίσει τι χώρε πρόέλευση και όχι τις χώρες εισόδου. τα χρήματα δεν έχουν σύνορα. τα κράτη όμω έχουν. αν συνεχίσετε να δίνετε βαρύτητα στα χρήματα θα εξαφανίσετε τα κράτη. αυτό επιδιώκετε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συναδεινέ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφο Κονσάλη Πόνς. Ευχαριστώ. Η αιτία της μετανάστευσης ε, είναι κυρίως η φτώχεια. Η μετανάστευση και η ανάπτυξη θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Το ξέρουμε γιατί ε, μεταναστεύσαμε πολλές φορές ε, για να επιτύχουμε ευημερία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έφτακτη μετανάστευση και ταυτόχρονα να αυξήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια από τις χώρες ε, προέλευση των μεταναστών. Το είπε και ο Ποντίφικας. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο, σε νεκροταφείο. Και γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να μην διακυβεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων, αλλά να προβλέψουμε μια αξιοπρεπή υποδοχή και φιλοξενία των μεταναστών. Η Ιταλία είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, δεν αρκούν μόνο περισσότερα χρήματα προς την Ιταλία αν δεν έχουμε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για την παράτυπη μετανάστευση. Η πατρίδα μου, η Ισπανία, είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ε, επίγειο χερσαίο σύνορο με την Αφρική. Και θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των, και την προστασία των συνόρων και την ασφάλεια των προσώπων που προσπαθούν να τα ξεπεράσουν. Δεν είναι ε, η καθημερινή αυτή διαχείριση εύκολη υπόθεση. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, η ρίζα του κακού είναι η φτώχεια. Εμείς προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Η μετανάστευση είναι απόρρια της φτώχειας. Η φτώχεια είναι η αιτία και ο αγώνας μας ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και όχι να στραφούμε κατά των μεταναστών. Θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να, κάνουμε τον αγώνα μας κατά της φτώχειας και όχι κατά των απόρων και των φτωχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέπετε ερώτηση του συνάδελφου Ουρτάσουν ε, με γαλάζια κάρτα. Επιτρέπετε μια ερώτηση του συναδέλφου, παρακαλώ. Δεν το βλέπω όμως που κάθεται. Μικρό. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Γκονσάλες Πόνς, πολύ ωραία αυτά που μας είπατε για την ανάγκη ενίσχυσης αναπτυξιακής συνεργασίας. Πώς το συνδυάζετε όμως αυτό με το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά μείωσε 7 ε, φορές την ε, βοήθειά της και τη συμβολή της στο Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης, συρρυκνώνοντας έτσι την αναπτυξιακή βοήθεια. Από τους μετανάστες που φτάνουν στα σύνορα της ΕΟΤΑ και της Μελίγες, ε, μόνο 5% ε, ζητούν άσυλο. Οι υπόλοιποι είναι οικονομικοί μετανάστες. Αν λοιπόν δεν διορθώσουμε τις οικονομικές αιτίες, δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη στη μετανάστευση. Θα πρέπει φυσικά να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια σε μια όμως κοινή ευρωπαϊκή, ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Αν δεν έχουμε κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, καμία χώρα από μόνη της δεν θα μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Ούτε η Ισπανία μόνη της, ούτε και καμία άλλη χώρα μόνη της. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε γνωρίζουμε και έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι ε, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Αναγκάζονται οι πρόσφυγες να, φύγουν, να ξεφύγουν από πολέμους και από τη φτώχεια. Και ξανά και ξανά λέμε ότι δεν μπορεί να είναι ένα υγρό τάφο η Μεσόγειο. Αλλά τι κάνουμε, περιμένουμε την επόμενη τραγωδία πριν γίνει οτιδήποτε κάθε φορά. Κύριε Επίτροπε, ε, έχετε μια πάρα πολύ σοβαρή δοκιμή τώρα μπροστά σα. Μια νέα ε, πολιτική ασύλου και μετανάστευση καλείται να διαμορφώσετε, η οποία θα αξίζει το όνομά τη και θα είναι στραμμένη προ το μέλλον. Γι' αυτό σα καλώ πραγματικά να ενισχύσετε τι προσπάθειέ σα για να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στην Ευρώπη για τη μετανάστευση. Μια πολιτική που πραγματικά να είναι και ανθρώπινη. Θα πρέπει να βρούμε έναν ασφαλή δρόμο για τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη, να τον εξασφαλίσουμε και να τους έχουμε και ένα μέλλον. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες ε, τα τελευταία 20 χρόνια τα θύματα. Το σύστημα ασύλου δεν λειτουργεί σωστά στην Ευρώπη. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο Πρόεδρος διακόπτη. Ε, η κυρία Φωνστόρχ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σήμερα μιλούμε για τη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για την πολιτική το πολιτικό άσυλο και τους πολιτικά διοκόμενους. Είπε ο Πάπας Φραγκίσκος το πρωί, δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, να γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο η Μεσόγειος και η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση εάν στις χώρες προέλευσης και καταγωγής βοηθήσει για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε τη ρίζα και όχι τις συνέπειες και ε, ο Σολ ε, Λατούρ, ε, ο συγγραφέας ο Γερμανός, είπε «Δεν μπορούμε να σώσουμε την Καλκούτα φέρνοντας όλη την Καλκούτα στην Ευρώπη». Δεν γίνεται αυτό. Είναι τεσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που πρέπει να ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια τη μέρα. Γι' αυτό έρχονται να πνιγούν στη Μεσόγειο. Είναι τραγωδία. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Στη χώρα τους πρέπει να βοηθηθούν οι άνθρωποι να έχουν ελπίδα. Ε, μόνο έτσι δεν θα αφήνουν τι οικογένειέ του, δεν θα μπαίνουν σε αυτά τα σαπιοκάραβα. Θα πρέπει να σώσουμε ζωέ, να βοηθήσουμε του φτωχού για να μην γίνονται οι φτωχοί μετανάστε τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φωνστόχ. Για ένα λεπτό η κυρία Βάινμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί ε, μπαίνουν ε, άνθρωποι σε σαπιοκάραβα διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από διωγμούς και πολέμους. Και είπατε αρμοστία των προσφύγων θα πρέπει επίσης να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης και φροντίζει για τους πρόσφυγες, αλλά ε, έχουμε ελεύθερη διακίνηση ε, με μερικές αφρικανικές χώρες. Έχουμε την οδηγία για τους εποχικά εργαζόμενους, και φυσικά επιτρέπουμε ένα βαθμό νόμιμη μετανάστευση, αλλά οι περισσότεροι μετανάστες ε, εξαπατώνται από τους διακινητέ και διακινδυνεύουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να αγνοούμε όλα αυτά τα προβλήματα και επίσης ε, τη λαθρεργασία. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για, για μια καλύτερη ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex δεν έχει βοηθήσει δυστυχώς ακόμη πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μάγερ για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ και ένα χρόνο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λαμπετούζας ένα πλοίο με εκατοντάδες ε, νεκρούς τελικά. Μάθαμε τίποτα, απάντηση όχι. Ε, συνεχίζεται η κατάσταση. Ε, οι κρατικές αρχές στην ε, Γαλλία και στην Ιταλία ε, δεν αντιμετωπίζουν την κατάσταση και εκατοντάδες ε, άνθρωποι που ζητούν άσυλο προωθούνται σε άλλες χώρες. Το Κοινοβούλιο ζητεί περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερα χρήματα και περισσότερους νόμιμους τρόπους να έρχονται οι μετανάστες στην Ένωση. Αλλιώς τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα. Εγώ είμαι από την Ολλανδία Έχουμε 29.000 ε, ε, ε, τούντες άσυλο και του χρόνου περιμένουμε και 40.000 αυξάνονται τα κέντρα υποδοχής, αυξάνονται οι δαπάνες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση, να κλείσουν τα σύνορα και να φροντίσουμε ε, να υπάρξει υποδοχή τους εκεί στην περιφέρεια. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τη μαζική μετανάστευση και τους θανάτους. Φοβούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε επιτόπου εκεί να βοηθηθούν στην περιοχή αυτοί οι άνθρωποι και να μην έρχονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μάιερ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Καρδίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς κάνουμε διαρκώς ε, λόγους γεμάτους ε, καλές προθέσεις ε, ε, οθούμενοι από τα, τις τραγωδίες που συμβαίνουν ε, στη Μεσόγειο. Ωστόσο, συγκεκριμένες απτές απαντήσεις, συγκεκριμένες απτές λύσεις δεν έχουμε δώσει. Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι η επιχείρηση τρίτων είναι το καλύτερο ή το χειρότερο για την Ιταλία. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι τέτοιου είδους λύσεις δεν μπορεί να είναι οι τελειωτικές λύσεις και δεν είναι ε, να χάνουμε από την άλλη μεριά τον έλεγχο των ε, συνόρων μας. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Το Μάρε Nostrum κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο δεν πέτυχε, αλλά είχε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Έχει σαν αποτέλεσμα αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών, έχει αυξηθεί το, το, το, ποσό των εσόδων των διακινητών που έχουν εκτραχυνθεί και κανένα αποτέλεσμα δεν είχαμε. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες χώρες οι οποίες ε, αποφασίζουν ε, να βοηθήσουν οικονομικά ωστόσο χωρίς να μπορούν να δώσουν τελειωτικές λύσεις. Και ο Πάπας το είπε σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να δράσουμε επί των αιτίων και όχι επί του αποτελέσματος. Θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες από τις οποίες οποίες προέρχονται οι μετανάστες όπως είπε και ο Ποντίφικας το πρωί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καρδίνη. Για ένα λεπτό κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τραγωδία της Λαμπεντούζα μας κινητοποίησε επιγόντως και εστιάσαμε την προσοχή μας στη Μεσόγειο. Υποδεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες. Διαπιστώσαμε όμως κενά στο μηχανισμό του Δουβλίνου και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί γιατί επιβαρύνει κυρίως τις χώρες που έχουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παραβιάζεται λοιπόν η αλληλεγγύη, δεν υπάρχει επιμερισμός των ευθυνών. Χρειαζόμαστε πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Τι γίνεται όμως με τα χερσαία σύνορα. Πρόσφατα βρήκαμε μετανάστες που είχαν παγώσει στα σύνορα Βουλγαρίας-Σερβίας. Τον Οκτώβριο 1.430 ε, άτομα πέρασαν τα σύνορα από την Τουρκία. Χρειαζόμαστε νόμι, νόμιμους ε, ε, δρόμους. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το, την εμπορία ανθρώπων, να ενισχύσουμε τη Frontex και να έχουμε κοινέ περιπολίες. Επίσης, να αποφύγουμε την εξαγωγή της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα. Το λόγο έχει η κυρία Στέβενση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκτός από την εμπιστοσύνη χρειάζεται συντονισμός και συνέπεια. Αυτά είναι για μένα οι λέξεις κλειδιά. Τώρα έχουμε κατακαιρματίσει τον προπολογισμό σε διάφορα ταμεία, σε διάφορες γραμμές, με ε, αυτό σκοπό το κάθε ένα και με ίδια γραφειοκρατική και διοικητική δομή. Λείπει η συνολική θεώρηση. Για τη μετανάστευση λοιπόν και το άσυλο είναι καλή αυτή η πρωτοβουλία και καλή εναλλακτική. Ε, δεν θα πρέπει ο κόσμος να μπαίνει σε περιπέτειες για να φτάσει στην Ευρώπη και θα πρέπει να σταματήσει ε, αυτή η ιστορία με τους διακινητές και τους δουλεμπόρους. Ε, ε, ε, η παράνομη μετανάστευση είναι αυτή που θα πρέπει να παταχθεί. Ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τι βήματα προτίθεται να αναλάβουν για να έχουν καλύτερο συντονισμό και εσωτερικό αλλά και εξωτερικό σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Στέβενς. Η κυρία Αρνοτού έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στη συνολική σας προσέγγιση ολιστική, λέει, της μετανάστευσης, ε, ο κύριος Μωράης αλλά και ο κύριος Αβραμόπουλος συστηματικά αποφεύγουν τα βασικά προβλήματα και δεν μας ε, καθησυχάζουν για το μέλλον. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία σε 12 κέντρα, από 12 κέντρα έχουν κλείσει τα 8 λόγω των εξεγέρσεων των παρανόμων. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, το είπε και ο κύριος Σαλβίνη. Οι Ιταλοί υφίστανται ε, την ε, ανάπτυξη 150-160 χιλιάδων παρανόμων στις ακτές τους μόνο το 14. Ε, παρά τα διάφορα που γίνονται για τα μάτια με τη Frontex και τα λεφτά, έχουν κάνει την Ιταλία σε ένα τεράστιο ε, κέντρο ε, διαλογής ε, πριν τους μοιράζουν στα διάφορα κράτη-μέλη Σέγγεν και μεταξύ αυτών και τη δική μου χώρα τη Γαλλία. Ε, εγώ ε, ε είμαι, εκλέγομαι στην Ίκαια που είναι κοντά στα σύνορα. Κάθε εβδομάδα έχουμε ε, ρεύματα πάνω από χίλιους. Ε, είπε λέει, το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να γίνουν ε, καλύτεροι χειρισμοί. Θα πρέπει αμέσως να αντιστραφεί αυτή η πολιτική, να διακοπεί, να ανασταλεί η συμφωνία Σέγγεν και να ανακτήσουν τον έλεγχο των σύνορων και την εθνική τους κυριαρχία τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αρναουτού. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Βόζεμπερκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επεσήμανα εγώ μια άλλη φράση στα λόγια του Άγιου Πατέρα το πρωί, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι το χαμένο βλέμμα των ανθρώπων αυτών ζητούν υποστήριξη και αποδοχή. Σήμερα στην πατρίδα μου, 30 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, βρίσκεται ένα καράβι ακυβέρνητο με 700 ψυχέ, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό από γυναίκε και μωρά. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν υποστήριξη και υποδοχή δεν, έχει καμία σημασία αν η χώρα μου είναι χώρα πρώτης υποδοχής χώρα διέλευσης ή χώρα τελικού προορισμού. σημασία έχει αν πράγματι στην πράξη στην ευρωπαϊκή ένωση γίνεται δίκαιη κατανομή αυτών που ζητούν άσυλο και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στην αλληλεγγύη η αλληλεγγύη φαίνεται ότι εξαρτάται και από συγκεκριμένα συμφέροντα. είμαι βέβαιη κύριε επίτροπε το επεσήμανα και στην εισήγησή σας ότι υπάρχει πράγματι η πολιτική βούληση να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς επίσης και να θεσπιστούν κανόνες για την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της ευρωπαϊκής ένωσης της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών που όπως γνωρίζετε αποτυπώνονται οι αρχές αυτές στο άρθρο 80 της σύμβασης για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης διότι πιστεύω ότι πρέπει όλα τα κράτη μέλη να αντιληφθούν ότι η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα είναι θέμα που αφορά σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ευρωπαϊκής ένωσης και επιπρόσθετα να επισημάνουμε ότι δεν νοείται με τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης να κατανέμετε η αλληλεγγύη σε δύο ή περισσότερες ταχύτητες. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βόζεμπεργκ και τώρα για ένα λεπτό η περισσοτερες ταχυτητες ευχαριστω πολυ ευχαριστω κυρια βοζεμπεργκ Γκυγιόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, οτιδήποτε σχετίζεται με την ε, μετανάστευση, όλες αυτές οι εκκλήσεις ε, μας δίνουν πληροφόρηση αλλά και παραπληροφόρηση. Πολλοί το είπαν πριν από μένα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε μία ευανάγνωστη βραχυπρόθεσμη πολιτική. Δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά με κοντόθωρες πολιτικές. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να είμαστε στρατευμένοι, δεσμευμένοι και με μια προενεργητική ε, ε, πολιτική. Ε, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, μια διαφορετική αντιμετώπιση εναλλακτική όλων αυτών που προσπαθούν να βρουν προστασία μέσω της μετανάστευσης. Σας άκουσα κύριε Επίτροπε πολύ προσεκτικά και σε πολλά σημεία συμφωνώ μαζί σας. Αλλά περιμένω με ανυπομονησία ουσία απτές συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα είναι άμεσες αλλά θα δρουν μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ κύριε Γκυγιώμα. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεταναστευτική πίεση θα αυξήσει. Η αιτία της ε, είναι η οικονομική διαφορά στο βιωτικό επίπεδο, αλλά και η καταβάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε χώρες που μαστίζονται από τους πολέμους και, την, και, τον, αυταρχισμό. Η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο περιζήτητος προορισμός. Ε, δεν θα πρέπει όμως να, επιτρέψουμε να γίνει μεγάλο ε, νεκροταφή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταναστευτικές ροές δημιουργούν προβλήματα αλλά και ευκαιρίες για την Ευρώπη, δημογραφικές και οικονομικές. Απαιτείται όμως μια περίπλοκη πολυσύνθετη μεταναστευτική πολιτική σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Εναρμόνιση των δραστηριοτήτων ώστε να μην μείνουν εγκαταλειμμένα στη μοίρα τους τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις δημογραφικές πιέσεις και στις μεταναστευτικές πιέσεις και να εξασφαλίσουμε και αξιοπρεπή ε, μεταχείριση των μεταναστών και των ετούντων άσυλο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, ε, τις εταιρικές μας σχέσεις με τις τρίτες χώρες, ε, να θεσπίσουμε προγράμματα επανεγκατάστασης. Ερωτώ λοιπόν, τι δράση αναλάβει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για να στηρίξει τα, τους μηχανισμούς πολιτικής γειτονίας, τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ώστε να μειωθεί η οικονομική ε, μεταναστευτική πίεση πώς ε, θα έχουμε αποτελεσματικό σύστημα ε, και μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πώς θα τηρήσουμε τις υψηλές προδιαγραφές του πακέτου μέτρων για το άσυλο, τι διορθώσεις θα πρέπει να κάνουμε στο σύστημα ώστε να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και να βοηθήσουμε την καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Είναι σημαντικό αυτό το διακόπτεται δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δεν βλέπω την κυρία Πόστο όμω και δίνω μέσω στο λόγο για 1,5 λεπτό στον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, κύριε ε, Υπουργέ Γκότσι, μετά το δράμα της ε, Λαπεντούζα άνοιξε τα μάτια της η Ευρώπη στο δράμα των μεταναστών και ε, χάρη στη δράση της ε, Ιταλικής κυβέρνησης περάσαμε από την προσέγγιση χώρας πρώτης υποδοχής σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ωστόσο, παραμένει το κατεπήγον του ζητήματος, όπως υπενθύμησε ο Πάπας Φραγκίσκος σήμερα το πρωί. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια Μεσόγειο που γίνεται νεκροταφείο. Πολλές είναι οι ανθρώπινες σοές ε, οι οποίες εισώθησαν ε, χάρη στο ε, Mare Nostrum. Συνεχίζει η Frontex, αλλά εγώ ρωτώ ποια είναι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την διεύρυνση της Frontex, ποια είναι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν τη διεύρυνση του προϋπολογισμού της Frontex, έτσι ώστε να υπάρξουν πολιτικές αποτελεσματικού ελέγχου στη Μεσόγειο. Ο τρίτον, κύριε Επίτροπε, δεν είναι η θα πρέπει ε, με θάρρος να αλλάξουμε πολιτική και θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσουμε τις ε, προσπάθειές μας στην αφρικανική ακτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε εκεί τις ε, καταστάσεις. Θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Γι' αυτό ζητούμε σήμερα δέσμευση και θάρρος έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και να περισσώσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ κύριε Λαβία. Λόπες Αγγιλάρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Επίτροπε, σε μία συζήτηση που δυστυχώ για πρώτη φορά γίνεται στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώ επειδή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Δεν θα είναι η τελευταία φορά όμω που θα έχουμε τέτοια συζήτηση, γιατί το συζητήσαμε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Όλοι λυπόμαστε για την έλλειψη τέτοια ολοκληρωμένη και κοινή πολιτική. Απαιτούμε την θέσπιση μια τέτοια πολιτική και αλλαγή τη εστίαση. Γιατί δεν είναι σωστή η εστίαση που έχουμε. Γιατί ουσιαστικά κλείνουμε τι πύλε στον στην νόμιμη μετανάστευση και εξωθούμε τον κόσμο στην παράτυπη μετανάστευση. Η Μεσόγειος έχει γίνει σε κάτι χειρότερο από υγρό από νεκροταφείο. Έχει γίνει ουσιαστικά ένα κοινό τάφος ε, μη αναγνωρισμένων πτωμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους και δεν μπορούν να βρουν δεκάν τα πτώματά τους. Θα πρέπει κατεπηγόντως να βρούμε μία απάντηση και να δώσουμε μία λύση. Και όχι μόνο για να απαντήσουμε στην τραγωδία της Λαμπεντούζα με μια επιχείρηση διάσωση στη θάλασσα που αμέσως ε, ε ακριβώς ε, προκάλεσε αντιδράσεις και αντικαταστήσαμε μία επιχείρηση με μία άλλη που δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα. Διακόπτει το μικρόφωνο του κ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Σέγγελ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στα ελληνικά ο κύριος Σέγγελ. Ε, έχουμε ως ε, εκπρόσωποι του λαού ε, το καθήκον να ενημερώνουμε σωστά την κοινή γνώμη. Ακούω διάφορα ανόητα, ε, στενόμυαλα και λαϊκιστικά από τη δεξιά και αισθάνομαι την ανάγκη να σας δώσω κάποια στοιχεία. 480 εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι μετανάστες απόδημοι και οι ε, κατιόντες συγγενείς τους. Ε, είναι όσος ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και λίγοι το έκαναν για λόγους ε, ευκολίας διασκέδασης ή ε, για να επωφεληθούν από την κοινωνική ασφάλιση. Και θέλω να πω στη νεαρή συνάδελφο από τις κάτω χώρες. Μας μιλάει για να κλείσουμε τα σύνορα, λέει, μα 15 εκατομμύρια είναι η απόδημη Ολλανδία ανά τον κόσμο με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Περισσότεροι από τους Ολλανδούς της Ολλανδίας είναι αυτοί, ξέρετε. Λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να ακολουθούμε και την αυτοαγιότητα αγιότητα το Πάπα που ήταν μαζί μας το πρωί, να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Η Ευρώπη είναι ε, μια ήπειρος αποδημίας πριν γίνει ήπειρος μετανάστευσης. Ο κόσμος χτυπάει την πόρτα μας, δεν έχουμε το δικαίωμα να τους την κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Αγγέλ και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Πύρη. Πρόεδρε. Πέρυσι Είχαμε αυτή την καταστροφή στη Λαμπεντούζα. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν απλό συμβάν επεισόδιο. Από την αρχή του έτους πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πνίγηκαν στη Μεσόγειο. Εκφράζω την ε, ελπίδα ο νέος Επίτροπος να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και να είναι μια ύψιστη προτεραιότητα και χαίρομαι γι' αυτό. Ένα χρόνο μετά ε, τι ε, καταστροφέ αυτέ στον όλεθρο τη Λαμπετούζα δεν έχουμε νόμιμο τρόπο να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ένωση. Χαίρομαι που το συζητάει ε, ο επίτροπο με τι χώρε για την αύξηση των ποσοστώσεων. Ε, είναι η μόνη νόμιμη οδό να μπει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω σύντομα να βρεθεί και μια συμφωνία για την ε, έκδοση ανθρωπιστική θεώρηση διαβατήριων. Επίση, οι χώρε τη Νότια Ευρώπη δεν συνεννοούνται με τι χώρε. Ε, ε, προορισμού στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ασυνεννοησία και να έχουμε μια κοινή πολιτική επιτέλους που να βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πύρη. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ανθρώπινε καταστροφέ και τραγωδίε ε, στη Μεσόγειο έδειξαν ότι δεν μπορεί η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική να αγκιστρώνεται σπασμωδικά στην προστασία των σύνορων. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία. Καταρχήν, για τη Frontex. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε το ρόλο της Frontex στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής προσέγγισης. Η επιχείρηση τρίτων περιορίζεται μόνο στον έλεγχο των συνόρων, γιατί είναι πενιχρός ο προϋπολογισμός της και ε, περιμένουμε τεχνικό εξοπλισμό από τα κράτη-μέλη έχουν με πολλές εκκρεμότητε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν για να συμπληρώσουν την επιχείρηση τρίτων στη Μεσόγειο. Επίση, θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα στο εμπόριο ανθρώπων και στο έργο των διακινητών. Έχουμε το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Ανθρώπων που έχουμε υπογράψει για την παράνομη διακίνηση και την καταπολέμηση τη Θα πρέπει ε, να εφαρμόσουμε το μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής του πρωτοκόλλου και να δίνουμε στοιχεία για τους διακινητές, για τους δρόμους, για τους τρόπους τελέχωσης και για τα πιο ευάλωτα και ευπαθή άτομα. Επίση, συνεργασία με τρίτε χώρε να καταπολεμήσουμε τα αίτια του κακού και της μετανάστευση πολιτικά και οικονομικά. Είναι προφανέ ότι η μεταναστευτική μα πολιτική θα πρέπει να είναι πλήρω ενταγμένη σε εξωτερικές μας δράσει, στις οικονομικές και εμπορικέ μα σχέσει στην πρόληψη των κρίσεων και των συγκρούσεων και στην αναπτυξιακή μα πολιτική. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συνεργαστείτε με την εκπρόσωπο Μογκερίνη, την ε, είπατε εκπρόσωπο και τον Επίτροπο Χάν για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ύψο των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα ε, είχαμε τις δύο τελευταίες ομιλίες που ζήτησαν βοήθεια διερμηνή, γιατί δεν γίνεται αυτή η ταχύτητα, δεν προλαβαίνουν να σας μεταφράζουν. Και εγώ θα δει, ε, διακόπτω τους ομιλητές στο εξή. Όταν είναι αυτές οι αστρονομικές ταχύτητες. Η συνάδελφος Λάιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Η Μεσόγειος είναι ευρωπαϊκή τράπεζα και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανοιχτό νεκροταφείο, πράγμα που είπε και σήμερα το πρωί ο ίδιος ο Πάπας. Ε, υπάρχουν Ευρωπαίοι οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους μετανάστες να πεθαίνουν, να πνίγονται ε, έτσι ώστε να αποθαρρύνονται οι υπόλοιποι να έρχονται. Ας μου το πούν αυτό ε, αυτοί που, που είδαν τα πτώματα στην Λαμπεντούζα. Η μόνη διαφορά ε, που δεν είχαμε πριν, δηλαδή τότε τα, πλοία, ε, ήταν ε, ότι πραγματικά δεν βλέπαμε τους νεκρούς και τους πνιγμένους. Και αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου, ότι υπάρχουν σήμερα στην Ολομέλεια άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να μην βλέπουν. Δεν είναι δυνατόν μία χώρα και μόνο όμως να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα πρέπει να ανοίξουμε ανθρωπιστικές διόδους. Θα πρέπει να μου πείτε κύριε Επίτροπε σας το ζητώ τι γίνεται με αυτήν την συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλάιν. μισή λεπτό ο συνάδελφος Πολιέζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε απόλυτη ε, ε, κατεπίγουσα κατάσταση αποτελεί η ε, μετανάστευση η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κυρίως στην αρχική φάση πλήρωσαν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες. Η επιχείρηση Mare Nostrum ε, ολοκληρώθηκε. Όπως είπε και η επικεφαλής της ομάδας μου ε, στην ουσία ε, οδήγησε σε, περισσότερες, σε περισσότερους μετανάστες και περισσότερες αφήξεις. Στα πρώτα στους πρώτους τέσσερις ε, ε, μήνες ε, του 2014 είχαμε αύξηση 800% ακριβώς δύο μήνες μετά την Mare Nostrum. Ευελπιστώ, αλλά αμφιβάλλω εάν η επιχείρηση τρίτων θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση. Ε, αυτό που θα έπρεπε είναι να αναμειχθούν και 27 χώρες, αλλά κυρίως να αλλάξει το Δουβλίνο 3. Εκεί που η χώρα της πρώτης υποδοχής αναλαμβάνει αποκλειστικά να δώσει ή όχι το δικαίωμα ασύλου. Θα πρέπει όλες οι χώρες να μπορούν να έχουν αυτήν την δυνατότητα Άλλωστε υπάρχει και σχετική ε, ε, απόφαση του δικαστηρίου η οποία εμέσως επιβεβαιώνει την προσέγγιση αυτή. Θα πρέπει χωρίς λαϊκισμούς και δημαγωγίες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την ασφάλεια των κρατών μελών με την αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουμε. Ευχαριστώ. λεπτό Grazie, Chair. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη στιγμή που συζητούμε το θέμα αυτό. Όχι επειδή επήγει ανάγκη ανάληψη δράση, αλλά και εξαιτία των πρόσφατων γεγονότων και τραγωδιών στη Μεσόγειο. Είναι εγκληματίες οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τη δυστυχία των ε, άλλων για να πλουτίσουν. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά τους ε, ε, Ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και παραπονιούνται για το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνεται καμία δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για τις εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Λιβύη, που η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να διαδραματίσουμε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο να συνεργαστούν τα κρατημέλη μεταξύ τους και να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη πολιτική, να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για να βοηθήσουμε τους μετανάστες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Κύρκος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα προσπαθήσω με τρεις λέξεις να περιγράψω το πρόβλημα. Η πρώτη είναι αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες που έρχονται από χώρες από ζώνες πολέμου και καταστροφών αλλά αλληλεγγύη και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Αλληλεγγύη με το ζόρι? Όχι. Αλλά ως Ευρωπαίοι περηφανευόμαστε ότι βρίσκουμε πάντα τρόπους για να συμφωνήσουμε. Εδώ είναι λοιπόν ένα πρόβλημα που πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεύτερη λέξη είναι κανόνες. Κανόνες για την νόμιμη οικονομική μετανάστευση. Κανόνες που παίρνουν υπόψη και τις φοβερές ανάγκες της γερασμένης μας υπήρου αλλά και τα όρια που μπορεί να ε, κρατήσει τα όρια των αναγκών της. Το τρίτο, η τρίτη λέξη είναι χρόνος. Χρόνος είναι κάτι που δεν έχουμε. Πολύ σωστά ο πρόεδρος Μωράς μας είπε ότι έχουμε τα εργαλεία. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μας διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή έχει τη θέληση. Αυτό που δεν έχουμε είναι χρόνος. Γι' αυτό από το Κοινοβούλιο θα μπορούσα να πω μόνο βιαστείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κύρκο. Ερχόμαστε στη διαδικασία Κατσιάη τώρα. Μόνο πέντε συναδέλφους ε, θα ακούσουμε. Ε, έχουμε πάρα πολλές αιτήσει, πολύ περισσότερες. Έλαβα υπόψη μου και τις πολιτικές ομάδες και τους έχω κόψει και το λόγο, ε, λόγω της πίσης χρόνου. Κύριο κύριος Κοέλιο πρώτος. Ευχαριστώ. Σχεδόν όλοι οι προλαλήσαντες μίλησαν για το ποντίφικα και το σχόλιο του ότι η Μεσόγειος δεν πρέπει να γίνει νεκροταφείο. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο έχουμε πολλά να κάνουμε. Κάτι όμως που μπορούμε να κάνουμε ήδη είναι να θέσουμε ως προτεραιότητα την διάσωση ζώων. Έχουμε εγκρίνει τον κανονισμό που δίνει προτεραιότητα στη διάσωση στις αποστολές της Frontex. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το καθήκον του. Το Συμβούλιο ήταν απρόθυμο στην αρχή αλλά τελικά υποχώρησε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί να αποφύγουμε την υποκρισία και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε δύο τινά. Πρώτον, να εφαρμόσουμε σωστά τον κανονισμό που εγκρίναμε και δεύτερον, να παρατείνουμε αυτές τις προτεραιότητες, τις διάσωσης δηλαδή και για τις αποστολές που είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνείτε μαζί μου κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέγιο. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή την πρώτη σας εμφάνιση έχω και εγώ την ευκαιρία να σας εκθέσω τις σκέψεις μου γύρω από το θέμα της παράνομης μετανάστευσης που όπως ξέρετε κυρίως χτυπάει τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου οι οποίες υποφέρουν έχουν φτωχοποιηθεί λόγω των μνημονίων λόγω της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν θα μείνω στο ζήτημα της αλληλεγγύης. πρέπει να υπάρχει κατανομή σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και αυτή η κατανομή θα πρέπει να έχει τρία στοιχεία να εξαρτάται από την έκταση από τον πληθυσμό και από το αεπ των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. η ελλάδα όπως ξέρετε δεν αντέχει άλλους παράνομους μετανάστες το ίδιο ισχύει και για την ιταλία. πρέπει ταυτόχρονα να τροποποιηθεί και το δουβλίνο 3 διότι δεν μπορεί η ελλάδα να μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Η κυρία Ντεσσαρνέζ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο χρειάζεται ε, ευρωπαϊκή απάντηση και αυτό είναι το θέμα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε οικοδομώντας μια κοινή πολιτική που θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, να υπάρχει πραγματική ασφάλεια και πραγματική προστασία και επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, διαθαλάσσεις, αέρος κλπ. Ε, το δεύτερο σημείο είναι επιστέγασμα του προηγουμένου. Θα πρέπει να ε, ε, ρυθμίσουμε την άδεια εισόδου ενδεχομένως μέσα από ένα αναχώρα. Τρίτον, είναι επίγουσα η κατάσταση και επίγει, το είπατε όλοι, να εναρμονίσουμε το δικαίωμα ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε καταστάσεις όπου σε μία χώρα μετά από πέντε μήνες παίρνεις άσυλο, σε άλλες μετά από πέντε χρόνια. Τέταρτος πυλώνας, μια πραγματική πολιτική συνεργασία συνεργασίας και ανάπτυξης με τις ε, χώρες ε, ε, από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύρια Δησανές. Ο κύριος Όμπεμάια παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα χρόνο μετά το μεγάλο ναυάγιο στη Λαβεδούζα και πάλι συζητάμε για ροές προσφύγων για συμπτώματα, δηλαδή δεν κοιτάμε τη ρίζα του κακού. Το Mare Nostrum ε, και το Τρίτον ε, είναι χρήσιμα, αλλά είναι απλή αντίδραση σε ε, μία μαζική άφηξη. Θα πρέπει να εκδημοκρατήσουμε τις περιοχές του κόσμου, να τις σταθεροποιήσουμε και να σταματήσει αυτή η αδίστακτη ε, λαιλασία των πρώτων υλών στις χώρες αυτές. Το είπε και ο Πάπας Φραγκίσκος. Ε, θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε τις συνθήκες πλαίσιο στις χώρες των ανθρώπων αυτών για να μην θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους. Βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποιοι ονειροπόλοι που το βλέπουν διαφορετικά, αλλά ε, δεν μπορούμε να φέρουμε και την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία ολόκληρη στην Ευρώπη. Δεν χωράνε. Ε, λοιπόν, να κάνουμε κάτι και οι πολίτες θα το εκτιμήσουν αυτό πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Ομπερμάιερ. Ε, να ολοκληρώσουμε η κυρία Μουσολίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι ούτε καν το ένα λεπτό. Έχουμε εδώ τον Υφυπουργό Κώση. Ε, το, οι περισσότεροι λένε οι περισσότεροι μετανάστες είναι παιδιά, είναι μικρά παιδιά τα οποία είναι κατατρομοκρατημένα. Το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια στην ε, Λαμπεντούζα και πρέπει να ε, τους δώσουμε ένα ε, πραγματικό νομικό καθεστώς γιατί δεν μπορούν να μείνουν απλοί αριθμοί. Οι αριθμοί χάνονται και γίνονται παιχνίδι στα χέρια των διακινητών. Θα πρέπει να τους δώσουμε λοιπόν ένα νομικό καθεστώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μουσολίνη. Εδώ ολοκληρώνεται και το Eye. Και για να κλείσει η συζήτηση έχει το λόγο ο Επίτροπος ο κύριος Αβραμόπουλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή ε, τις ερωτήσεις που τέθηκαν από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να οδηγηθώ καταρχήν σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές όλες και όλοι με ελάχιστες εξαιρέσεις συμφωνούμε ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό έχει κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις και δοκιμάζει καθημερινά τις αρχές πάνω στις οποίες γεννήθηκε και θεμελιώθηκε η ευρώπη. δεν είμαι εδώ για να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση δεν έχω αυτή την πρόθεση. μπορεί να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση μονάχα τρεις εβδομάδες αλλά γνωρίζω και βιώνω το πρόβλημα από κοντά για πάρα πολλέ δεκαετίε και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσωπική αναφορά λέγοντα ότι όταν πριν από δεκαοκτώ περίπου χρόνια τα πρώτα κύματα παράτυπων μεταναστών χτυπούσαν τι πόρτε τη ευρώπη ήμουν δήμαρχο τη πόλεως των αθηνών και δεν κρύβω ότι ευνηδιάστηκα. ευνηδιάστηκε μαζί μου και το κράτο όπω ευνηδιάστηκαν και όλα τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου όταν άρχισαν να χτυπούν την πόρτα τη ευρώπη όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που ζητώντας μια καλύτερη θέση στον ήλιο και στη ζωή και σπρωγμένοι από τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπιζαν και που είχαν να κάνουν και με τη φτώχεια και με τον πόλεμο και με τις τραγωδίες που συνοδεύουν το προσωπικό τους δράμα. αναφερθήκατε στη Λαπεντούζα που έγινε σύμβολο για ολόκληρη την ευρώπη. δεν είναι μονάχα η Λαπεντούζα. εκεί θρηνήσαμε ανθρώπους την άλλη μεριά εκείνοι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας πούν που βρίσκονται γιατί χάθηκαν στα βάθη της μεσογείου και είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής από τα κράτη μέλη της ευρύτερης περιοχής. αγαπητοί ευρωβουλευτέ πολλοί πίστευαν στην αρχή ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα που αφορούσε στον ευρωπαϊκό νότο για να εξελιχθεί μέσα σε λίγα χρόνια στο να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ολόκληρης της ευρώπης. είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. πρέπει όμως να ξεχνάμε κάτι και αυτό για να απαντήσουμε σε όλους εκείνους που καλλιεργούν την ξενοφοβία και που δυστυχώς ξεθεμελιώνουν τις αρχές και τις αξίες ή τουλάχιστον το προσπαθούν πάνω στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. ότι όπως είπε ο κύριος Σέγγελ θα συμφωνήσω μαζί του είμαστε μια ένωση λαών και εθνών που όλοι εμείς ή τουλάχιστον οι προγονείς μας έστειλαν εκατομμύρια συμπατριωτών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. μεγάλες χώρες υπερδυνάμεις σήμερα είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων όπου κυριαρχεί το ευρωπαϊκό στοιχείο και οι δικοί μας άνθρωποι τότε ανάμεσά τους και συγγενείς μας παππούδες μας ή και παραπέρα αντιμετωπίστηκαν σκαιότατα. αντιμετωπίστηκαν με ξενοφοβία και με ρατσισμό τα έχει βιώσει λοιπόν αυτά ο ευρωπαίος πολίτης και έρχεται σήμερα μπροστά στις αξίες τις δικές του να δοκιμαστεί. πώς όμως; όχι με μια κατακαιρματισμένη πολιτική ούτε να τα φορτώνει ο ένας τον άλλον γιατί ακούστηκαν και τέτοιες φωνές εδώ μέσα αλλά για μια ολιστική συγκροτημένη στρατηγική μετανάστευση. υπάρχει ναι σας διαβεβαιώνω το είπα και στο ξεκίνημα της σημερινής μας συζήτησης η πολιτική βούληση η επιτροπή είναι αποφασισμένη να υιοθετήσει μια νέα χάρτα για τη μετανάστευση γιατί αγαπητές και αγαπητοί ευρωβουλευτές το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε ή το ζήτημα θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξεπεραστεί. γνωρίζετε πώς εξελίσσονται γεωπολιτικά τα πράγματα σε όλο αυτό το τόξο αστάθειας που ξεκινά την τινησία και φτάνει στην ουκρανία. αυτή τη στιγμή στις ακτές της τουρκίας της λιβύης της αιγύπτου ή και αλλού βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που περιμένουν να βρουν έναν τρόπο να περάσουν απέναντι και είναι θύματα και των smugglers και των traffickers και όλων αυτών που όπως σας είπα πρωτήτερα είμαστε αποφασισμένοι σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να τους χτυπήσουμε αλίπητα. υπάρχουν χώρες ανάμεσα σε εκείνες και η ελλάδα από όπου προέρχομαι που ήδη πήραν πολύ αυστηρά μέτρα. τα ισόβια είναι μια ποινή που επιβάλλεται από τα δικαστήρια αυτής της χώρας και μην ακούσω όλους εκείνους που ξαφνικά θυμούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των smugglers. δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ξεπουλούν τις ανθρώπινες ψυχές γιατί πίσω από όλα αυτά που συζητούμε σήμερα εδώ κρύβεται πλέον και λειτουργεί μια τέλεια βιομηχανία εξοπλισμένη με τα καλύτερα συστήματα με νέες τεχνολογίες σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα εξοπλισμένη και οργανωμένη από τα ίδια τα κράτη. αντέδρασε η ευρώπη η πολιτική την οποία σήμερα επικρίνουμε είναι τον χρόνο που πέρασε είχε αρχίσει να δίνει αποτελέσματα. δοκιμάστηκαν κάποια προγράμματα. όπου αυτά απέτυχαν σταματούν. Καινούργια όμως προτείνονται. εμείς στηρίζουμε τα κράτη μέλη στις πολιτικές που αναλαμβάνουν. αλλά τώρα δεν θα είναι μόνα τους. το είπα πρόσφατα σε συναδέλφους πολιτικούς από τις χώρες κυρίως του ευρωπαϊκού νότου ότι οι χώρες τους δεν είναι μόνες είναι η ευρώπη κοντά τους και η ευρώπη θα αντιδείξει στην πράξη την αλληλεγγύη κυρία βόζεμπεργκ είναι υποχρέωσή της είναι μια από τις αρχές πάνω στι οποίε στηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και δοκιμάζεται καθημερινά και σε ζητήματα κοινωνικά ανθρωπιστικά πολιτικά. εδώ σε αυτόν τον ιερό χώρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που είναι ο ναός της ευρωπαϊκής δημοκρατίας όλες αυτές οι αρχές καθημερινά δοκιμάζονται και μέσα στι δικέ σας συζητήσεις. η επιτροπή έχει ανάγκη τη βοήθειά σας τη στήριξή σας τις ιδέες σας και τις ευαισθησίες σας ευαισθησίες που μοιραζόμαστε όλοι ανεξάρτητα σε ποιο θεσμικό όργανο της ευρώπης και αν βρισκόμαστε. εκείνο το οποίο μπορώ εγώ σήμερα να σας πω διότι όλα όσα ελέγξαν πρωτήτερα είναι προς την ίδια κατεύθυνση η οποία σας το επαναλαμβάνω έχει να κάνει με τη βούλησή μας να υιοθετήσουμε μια νέα χάρτα για τη μετανάστευση που θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και όλε τι ανθρωπιστικέ αξίε και αρχέ που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον τόπο που λέγεται ευρώπη και που δίνουν σήμερα στον κόσμο ολόκληρο το λαμπρότερο παράδειγμα της δημοκρατίας στην πράξη. γι' αυτό η ευρώπη είναι ελκυστική και γιατί ευημερεί και γιατί εδώ γνωρίζει ο άλλος ότι θα τον σεβαστούν. ξέρουμε που πάσχει το σύστημα. γνωρίζουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του διότι η εμπειρία που αποκόμισε η προηγούμενη επιτροπή αλλά και όλοι εσείς εδώ μέσα πέρασε σε εμάς και μεταφράζεται στην απόλυτη ευθύνη να υιοθετήσουμε πλέον μια συγκροτημένη ολοκληρωμένη πολιτική που θα απαντάει στο ζήτημα με ευαισθησία ανθρωπιά που θα αναδεικνύει αρχές και αξίες που δοκιμάζονται στην πράξη και που ναι σε κάποια στιγμή όλοι μαζί θα αποφασίσουμε να ξεκαθαρίσουμε την έννοια των ευρωπαϊκών συνόρων. αλλά τα σύνορά μας δεν θα οδηγήσουν ποτέ το χαπί αν θυμόσαστε και στο hearing στην ακρόαση που πέρασα μπροστά σας σε αυτό που ήταν σύνθημα του μεσοπολέμου και ξέρετε από ποιους προερχόταν αυτό το σύνθημα δεν αξίζει ούτε να τους ονοματίσω σε αυτή την αίθουσα για μια ευρώπη φρούριο. Ε, λοιπόν, η Ευρώπη δεν θα γίνει φρούριο, η Ευρώπη δεν θα οδηγηθεί στον απομονωτισμό, η Ευρώπη αποτελείται από πολίτες του κόσμου και έχει ανοιχτέ ακριβώς τις πόρτες της στους άλλους πολίτες του κόσμου που οι δύσκολες καταστάσεις τους οδήγησαν κοντά μας σήμερα αναζητώντας μια καλύτερη υποδοχή πιο ανθρώπινη ένα καλύτερο πιο ανθρώπινο περιβάλλον και δυνατότητες να ασκήσουν κοντά μας το δικαίωμά τους στη ζωή. αλλά όλα αυτά πλέον οργανωμένα κάτω από ένα πλέγμα αρχών αξιών και οδηγιών που θα εκπορεθούν μέσα από τη δική μας συνεργασία από αυτόν τον χώρο. αυτή τη διαβεβαίωση εγώ σήμερα θα ήθελα να σας δώσω ότι η ευρώπη των αξιών θα κριθεί στην πράξη η ευρώπη θα μπορέσει να ορθώσει το ανάστημά τη σε όλα αυτά που περιγράψαμε πρωτήτερα με πρώτο εκείνο που έχει να κάνει την εκμετάλλευση του ανθρώπου και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα αργήσει η μέρα που όλοι μαζί θα ζήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. εύχομαι πραγματικά με την καρδιά μου στο τέλος του επόμενου χρόνου να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις γιατί θα κάνουμε πολλές και ο σάκης μεγαλύτερη θα είμαι παρόν σε κάθε παρόμοιο ζήτημα αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε να έχουμε κάνει το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και προς τα πάνω δίνοντας πραγματικά απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα και να μην διονύζεται μια κατάσταση η οποία στην τελευταία ανάλυση προσβάλλει και εμάς και τις αξίες πάνω στις οποίες έχουμε θεμελιώσει το κοινό ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Βραμόπουλε. Και τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου ο Υπουργός κ. Γκόζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο σήμερα σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν είναι νέα συζήτηση βέβαια αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό που λαμβάνει η χώρα στην αρχή της ε, νέας κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Ε, σε αυτόν τον νέο πολιτικό κύκλο υπόθηκε άλλωστε θα πρέπει η Ευρώπη να ξεκινήσει με, με δύναμη γιατί διαφορετικά θα υπολείπεται διαρκώς και θα, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα τεστ αντοχής τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Χρειάζεται όπως είπαμε ολοκληρωμένη προσέγγιση πολλοί μεταξύ ημών ε, ε, είπαν ε, και το συμμεριζόμαστε εμείς σαν Προεδρία ότι θα πρέπει δηλαδή να συνδυαστούν οι εξωτερικές και οι εσωτερικές πτυχές, εξωτερική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική ε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν ε, οι μετανάστες. Ε, ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να προσέξουμε την πτυχή της ασφάλειας και να μπορέσουμε σιγά σιγά να φτάσουμε ενδεχομένως σε μια ευρωπαϊκή αστυνόμευση των συνόρων. Γενικά δουλεύουμε προς όλες αυτές τις οδούς και προς όλες αυτές τις διαδικασίες και εμείς Συμβούλιο λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, συνεργαστούμε με τις χώρες ε, προέλευσης, με τις χώρες διαμετακόμισης ε, και να εργαστούμε με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και να βελτιώσουμε και την πολιτική επιστροφή στις χώρες προέλευσης συνεργαζόμενοι οπωσδήποτε και με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες ε, όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της ε, μεγαλύτερης συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αναφερθήκατε στις διασώσεις στη θάλασσα. Υπενθυμίζω ότι η διάσωση οποιοδήποτε η ζωή του κινδυνεύει στη θάλασσα είναι διεθνής υποχρέωση, απορρέει από τις διεθνείς συνθήκες. Πρέπει να σώζονται οι άνθρωποι αυτοί ανεξάρτητα από την την υπηκότητά τους και εγώ θα προσθέσω ανεξάρτητα από το καθεστώς, από το στάτους ε, που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, να μελετήσουμε, να ελέγξουμε εκείνη την ώρα που πνίγεται κάποιος εάν θα ζητήσει άσυλο, αν έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο, εάν είναι οικονομικός μετανάστης κτλ. Θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, υπάρξουν ε, κοινέ επιχειρήσεις όπως η Frontex ή όπως ο Τρίτονας. Η επιχείρηση Τρίτον βεβαίως είναι μια αρχή, δεν αποτελεί τέλος. Νομίζω ότι αποτελεί μια καλή βάση, ένα καλό σημείο εκκίνησης. Βεβαίως θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και βεβαίως χρειάζονται περισσότεροι πόροι στην ε, νέα θητεία ε, και του ε, Συμβουλίου και εκεί έχει αναγνωριστεί η ανάγκη κοινή αντιμετώπισης. Αλλά βεβαίως και το τονίζω και το υπογραμμίζω χρειάζεται αλληλεγγύη και χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εάν μεταξύ μας δεν οικοδομήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, ό,τι και να κάνουμε θα παραμείνει κενό γράμμα. Ό,τι και να αποφασίσουμε θα παραμείνει στα χαρτιά γιατί ε, στην ουσία ε, από τη μία έχουμε χώρες ε, οι οποίες λένε ότι είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των ετούντων άσυλο. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες φτάνουν ανεξέλεγκτοι αριθμοί μεταναστών και λένε ότι δεν μπορούν να τους απορροφήσουν. Πολύ συχνά τίθεται ένα εσφαλμένο ερώτημα σχετικά με το ποιος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, ο ένας ή ο άλλος. Αυτός που δίνει περισσότερες άδειες, αυτός ε, που υποδέχεται περισσότερους μετανάστες. Ε, αυτό είναι ένα εσφαλμένο ε, ερώτημα. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε και τις δύο περιπτώσεις. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις η μόνη δυνατή απάντηση είναι μία νέα πολιτική, μία νέα αντιμετώπιση και δεν είναι δυνατόν ε, να μπούμε σε ένα παιχνίδι του ποιο έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μα μια πολιτική την οποία θα πρέπει να οικοδομήσουμε βήμα το βήμα και πρόταση την πρόταση. Το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ε, εξεπώνησε μια νέα οδηγία ε, και αυτό είναι μια ψηφίδα που αφορά την, την την άδεια ε, εγκατάστασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ερευνητών, επιστημόνων κτλ. Ε, σιγά σιγά θα προσθεθούν και άλλες ε, ψηφίδες. Θα υπάρξει και μια πρόταση ενδεχομένως της Επιτροπής σχετικά με την σωστότερη κατανομή του άχθους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε επίσης και εγώ το ανέφερα στην εισαγωγή μου συνόδευτη ανήλικη. Οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να ε, μελετήσουμε όλα τα όρια και τα περιθώρια τα οποία ε, μας ε, παρέχονται από το Δουβλίνο έτσι ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικότερα να δουλέψουμε. Υπενθυμίζω ότι ήδη πολλές χώρες δουλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή. Το συζητήσαμε άλλωστε και στις εργασίες του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να απαντήσω σε όλες τις παρεμβάσεις, αλλά ε, είναι γεγονός ότι ή θα πρέπει να δείξουμε τη βούληση ε, και το θάρρος ε, και την εμπιστοσύνη για να αντιμετωπίσουμε με κοινού τρόπους το πρόβλημα αυτό ή διαφορετικά θα αποτύχουμε σαν Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με την τοποθέτηση του Υπουργού ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα γίνει ε, στην επόμενη ε, σύνοδο. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα στη μέρη διάταξη που είναι προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και προτινόμενη νομιμοποίηση των εξαναγκαστικών επιστροφών στην Ισπανία. Πέντε ε, είναι οι συντάκτριες.